Good morning, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Uh, Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση. Υπάρχουν σχόλια? Όχι. Σημείο 2. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι δεν έχω ανακοινώσεις. Περνάμε τώρα στο σημείο 3 του τέστην έκθεση πρόοδου για το 2015 για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για πρώτη φορά θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης για τη Μακεδονία. Το 2015 η χώρα αυτή αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις και από και από διεθνείς εξελίξεις, ε, ασκώντας πίεση στην ε, σταθερότητά της. Καταρχήν εσωτερικά ε, ξέσπασαν κάποια σκάνδαλα υποκλοπών. Αυτό αποκάλυψε ο αρχηγός αντιπολίτευσης, κάτι που οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Δημιουργήθηκε μια πόλωση και έντονες πολιτικές εντάσεις μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης, κάτι που απείλησε την εσωτερική ισορροπή και σταθερότητα της χώρας. Τελικά συνήθει η τετραμερή συμφωνία τον Ιούνιο και Ιούλιο υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Διεύρυνσης και τριών μελών της Επιτροπής μας και χαίρομαι γι' αυτό οι ε, κύριοι Κούκαν, Χαουίτ και Βάγκλ ήταν οι τρεις ευρωβουλευτές που συμμετείχαν. Τώρα θα πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες ε, με βιώσιμο τρόπο από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεύτερον, φέτος η χώρα αντιμετώπισε πρωτοφανή ροή προσφύγων που διέσχισαν τη χώρα Μάλιστα η χώρα αντέδρασε ως υπεύθυνο εταίρος και προσπάθησε να διαχειριστεί τη διέλευση περίπου μισού εκατομμυρίου προσφύγων. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, διευκολύνει τις ε, δυνατότητες ε, υποδοχής και φιλοξενίας και να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο τα σύνορά της. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέκτηνε την σύσταση στο Συμβούλιο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαιτία των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα και εξαιτία τη μη τήρηση των ανηλυμένων υποχρεώσεων τη Συμφωνία Ιουνίου και Ιουλίου. Μετά τι 24 Απριλίου θα επανέλθει η Επιτροπή στο θέμα αυτό, τότε που θα γίνουν και οι πρόορε εκλογέ στη χώρα. Ο μόνιμο ηγητή μα για την ΕΦΙΡΟΜ είναι ο κύριο Βάγκλ, που αναλύει τα σχετικά με την ένταξη, ε, την πόλωση που έχει δημιουργηθεί, την πολιτικοποιημένη δικαστική εξουσία, τη δημόσια διοίκηση, ε, την κοινωνία των πολιτών, μια επαναχώρηση που έγινε σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και άλλα θέματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας. Αυτά και θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ιβο Βάγκλ, για μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσής του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, δηλαδή τα σλοβενικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Ως ε, εισηγητής για τη Μακεδονία φέτος, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η χώρα αυτή να προχωρήσει στρατηγικά και να γίνει και μέλος των Ευρωατλαντικών Συμμαχιών. Θέλουμε να μπορέσει να κάνει τα πρώτα επίσημα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και να μπορέσει να συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια καθώς και την πρόοδο της γενικότερης ευρωπαϊκής επικράτειας, της οποίας αποτελεί μέρος. Τους τελευταίους μήνες ξέρουμε ότι πέρασαν από τα Βαλκάνια εκατομμύρια πρόσφυγες ετούντες άσυλο και μετανάστες, οι οποίοι αναζητούν που μπορούν να ζήσουν καλύτερα ε, και προστατευμένοι. Είναι γεγονός ότι η Μακεδονία είναι μία από τις χώρες κλειδιά για τα Βαλκάνια με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η ίδια η χώρα, όπως ε, την πολυπολιτισμικότητα και τις, ε, τις διαφορετικές θρησκευτικές ε, μειονότητες. Εδώ λοιπόν η χώρα αυτή πέρασε από πολιτική κρίση, από καχυποψία έναντι των πολιτικών ηθινόντων, από κοινοβουλευτική κρίση και υπήρξαν και διάφορες συλλήψεις και υποκλοπές που έδειξαν ότι υπήρξαν πολλές καταχρήσεις και παραβιάσεις. Και επίσης και μια τρομοκρατική διάσταση. Ε, είδαμε σήμερα ότι στα πολιτικά πράγματα της ε, Μακεδονίας επικράτησε η λογική και η υπευθυνότητα έναντι των εσωτερικών της χώρας. Η συμφωνία που επετέφθη με τον Επίτροπο Χάν και τρία μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Μακεδονίας οδηγεί τη χώρα σε μια νέα περίοδο βάσει ε, των, συμφωνιών του 2 της Δευτέρας Ιουνίου 2015 Έχουμε πλέον μια κυβέρνηση σωστά διαφρομένη, έχει διοριστεί και υπουργό Εσωτερικών για να παρακολουθήσει το θέμα των υποκλοπών, των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχουν προβλεφθεί νέες θέσεις ελέγχου στο Κοινοβούλιο για την λογοδοσία της κυβέρνησης και έχει αποφασιστεί και η ημερομηνία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου. Το ψήφισμα αυτό επικεντρώνεται στα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την προσχώρηση της ε, Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει του ψηφίσματος για το οποίο σίγουρα θα υποβληθούν πολλές τροπολογίες, εντοπίζουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ήδη η χώρα από χρόνια έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχει ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, από την άποψη την εμπορική έχει πολύ καλή οικονομική ανάπτυξη, συνεργάζεται με τρόπο αποτελεσματικό στις αποστολές στήρησης της ειρήνης, αλλά υπάρχουν και επικριτικά σχόλια. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχει μεγάλη πολιτική πίεση προ τα μέσα μαζική ενημέρωση. Η χώρα δεν είναι έτοιμη να συνεργαστεί επαρκώ ε, στου επίσημου φορεί, στο επίπεδο των επίσημων φορέων με την κοινωνία των πολιτών. Επίση χρειάζεται μεταρρύθμιση στο δικαστικό τομέα. Και υπάρχουν μια σειρά από μεταρρυθμίσει που είναι απαραίτητε στη, χώρα αυτή. Στηρίζει όμω η Μακεδονία τη στήριξή μα στην πορεία της προς την ένταξή της στις ευρωτρατικές συμμαχίες. Τα προβλήματα που παραμένουν στη χώρα αυτή δεν θα έπρεπε να επηρεάσουν ή να ε, παρεμποδίσουν τη διαδικασία προσχώρησής της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η είπατε πρόσωπος, ε, η κυρία Μογκερίνη, θα πρέπει να πιέσει περισσότερο και να επηρεάσει στην ε, άρση όλων αυτών των φραγμών που δυσκολεύουν την πρόοδο της χώρας. Θα χρειαστεί διμερή συμφωνία για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να ανοίξει ο δρόμος για μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ γειτονικών χωρών. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να στηρίξετε αυτήν την θετική μας αποτίμηση προς την Μακεδονία και τον λαό της. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κυρία Μαριάννα Πετήρ που αντικαθιστά εδώ τον κύριο Πέτερλε που είναι ο πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπής για τις σχέσεις με τη Μακεδονία. κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα εκ μέρους του κυρίου Πέτερλε που δυστυχώς κολλείεται σήμερα και που είναι πρόεδρος ε, της ε, και ηγήθηκε της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μετέβη στη Μακεδονία και είναι και ο πρόεδρος, όπως είπατε, της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπής για τις σχέσεις με τη ΦΥΡΟΜ. Είχαμε μία πολύ καρποφόρα και πολύ δυναμική συνάντηση στην Βουλή με τους ε, ομολόγους μας της Μακεδονίας. Μετά την επιστροφή της αντιπολίτευσης ε, στη Βουλή ξαναξεκίνησε ο διάλογος ε, και για εκρεμή ζητήματα Ιδιαίτερα επικεντρωθήκαμε στο θέμα του κράτους δικαίου, ε, της δικαστικής εξουσίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, το θέμα της Επιτροπής, ε, Εθνικής Επιτροπής Εκλογής, ε, το θέμα της ελευθεροτυπίας και φυσικά την προσφυγική κρίση. Μετά τις συζητήσεις καταλήξαμε και σε κοινή διακήρυξη με μια σειρά συστάσεων και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών αλλά και των βουλευτών της ΦΥΡΟΜ ε, τάχθηκαν υπέρ αυτής της διακήρυξης με, εξαίρε, με εξαίρεση την επιφύλακτη, με την αποχή ε, του Έλληνα και ε, μία εποχή Έλληνα και οι υπόλοιποι Έλληνες ήταν κατά. Ε, και από τις συζητήσεις ότι η Μακεδονία πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο και αυτή η δεκαετής αναμονή δεν είναι δίκαιη για τη Μακεδονία, ούτε για την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ούτε και για την Μακεδονική Βουλή. Η βασική ε, πολιτική συμφωνία που ε, υλοποιήθηκε τον Ιούλιο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα της Μακεδονίας και ανοίγει πάλι το δρόμο της προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο της κρίσης. Γιατί στις εκλογές αναδεικνύεται η εξουσία και έγιναν πέρυσι εκλογές στη Μακεδονία. Η αντιπολίτευση προκάλεσε αυτή την κρίση, κάτι που επιβράδυνε τις μεταρρυθμίσεις, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και δεν νομίζω ότι η Μακεδονία αξίζει να περιμένει ούτε και μία μέρα ακόμη, να μην, να μην μείνει χαμένη ούτε μία μέρα. Μάλιστα ήταν αποθαρρυντική η κατάσταση αυτή ε, για την Μακεδονία και πιστεύω ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να στηρίξουν αμέριστα τη χώρα αυτή. Γιατί έχει πάρα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολύ δύσκολο έργο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρεται πολύ συχνά όταν μιλούμε για τη Μακεδονία. Θα πρέπει να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις και τη διμερή αντιπαράθεση που υπάρχει θα πρέπει να την αφήσουμε κατά μέρου και να επιληθεί με βάση την κοινωτική νομοθεσία. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έλυσαν τα διμερεί προβλήματα η Σλοβενία και η Κροατία είναι παράδειγμα προς μίμηση και για τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα με τη Μακεδονία. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειες της μακεδονικής κυβέρνησης που προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίσει το κράτος δικαίου και να προωθήσει αποτελεσματικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και τη διαφθορά. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Σας είπαμε σύντομη παρέμβαση κυρία Πετήρ. Ελάτε παρακαλώ στο διατάφτα. Μάλιστα. Εκ μέρου λοιπόν και του συναδέλφου Πέτερλε και της αντιπροσωπείας μας αλλά και εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε πως η Μακεδονία θα πρέπει και επίσημα να ξεκινήσει τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την αίτηση της Μακεδονίας για ένταξη και στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στους κοιόδους εισηγητές και στους ε, ενδιαφερόμενους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Κούκαν πρώτα. Ε, Θα σας δώσω την παρέμβαση του κυρίου Κέλλαν, τη σύντομη εκδοχή, που είναι ο εισηγητής για το ΕΛΚ. Θετική αποτίμηση για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για προσχώρηση της χώρας, η οποία περιμένει εδώ και πολύ καιρό και πλέον εκπληρώνει τη συμφωνία του καλοκαιριού ως προς την, τις μεταρρυθμίσεις στην, ε, και εάν υπάρξει και επιτυχή διοργάνωση των εκλογών μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι υψηλού επίπεδου και η ευθυγράμμιση της χώρας με το κεκτημένο. Το και επενεί τη χώρα για την πρόοδο στις συμφωνίες του φετινού Ιουλίου και Ιουνίου και η κυβέρνηση έχει δείξει ότι έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της περνώντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και νόμους. Η τεχνοκρατική κυβέρνηση που έχει αναλάβει, η υπηρεσιακή κυβέρνηση που έχει αναλάβει ρόλο τώρα, ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε επιτυχή διοργάνωση εκλογών την άνοιξη του 2016 στις 24 Απριλίου ακριβώς. Ε, δίκες και ανεξάρτητες εκλογές εφαρμόζοντας την συμφωνία. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία γιατί είναι σημαντικό μια χώρα μικρού να είναι δύσκολο εύκολο μάλλον μια τέτοια μικρή χώρα να αντιμετωπίσει μόνη τη την κρίση των προσφύγων. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ενταθούν οι προσπάθειε ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για τη ΦΥΡΟΜ. Ε, Επίση είναι και πολύ αρνητικέ οι συνέπειε στην οικονομία τη χώρα από την παρουσία των προσφύγων. Ο ειδικό εισαγγελέα θα πρέπει να διεξάγει ανεξάρτητε έρευνε για την περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Θα πρέπει να υπάρξει συστηματική καταπολέμηση τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει την τεχνογνωσία και τις απαραίτητες ε, δομές αρρωγής, συνδρομής σε όλα τα επίπεδα. Στην κυβέρνηση, την υπηρεσία και κυβέρνηση τώρα και στο μέλλον, καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία με τη κοινωνία των πολιτών. Αυτά λέει ο κύριος Κέλλαν, ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πιτσούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Βάγκλ για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Ε, μας παρέθεσε όλες τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει σήμερα η Μακεδονία. Ένα ολόκληρο φάσμα. Για παράδειγμα, εκλογική μεταρρύθμιση και επικείμενε πρόορες εκλογέ. Λυπούμε από καθυστέρηση η εκλογική μεταρρύθμιση και κυρίω σε ό,τι αφορά την επιλογή των μελών τη ε, Εθνική Εκλογική επιτροπή. Ελπίζω να ολοκληρωθεί η σύνθεση αυτής της Επιτροπής το συντομότερο δυνατό με συμμετοχή ανεξάρτητων επιρρογνωμόνων, ώστε να μην έχει κομματικό χαρακτήρα. Επίσης, ε, καλό για κατεπίκουσες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στη Μακεδονία σε σχέση με τον ε, κατάλογο, τους εκλογικούς καταλόγους. Γιατί είχαμε πολλές περιπτώσεις πλαστών ε, ταυτοτήτων και διαβατηρίων και πολλές ανακρίβειες στους ε, καταλόγους των ψηφοφόρων, κάτι που δημιούργησε πρόβλημα στην εκλογική διαδικασία, όπως φαίνεται και σε προηγούμενες ε, εκθέσεις της ΟΑΣΕ θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των εκλογών. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις 52% των πολιτών θεωρούν ότι οι κρατικοί θεσμοί ε, δεν είναι ικανοί, δεν είναι δεόντως ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ε, της εκλογικής αναμέτρησης. 44% ε, δεν πιστεύουν καν ότι είναι αξιόπιστη η εκλογική κατάλογη. Τέλος, ε, θεωρώ ότι η εκλογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της όλης διαδικασίας που θα διηγήσουν την Μακεδονία μακριά από την αποτελμάτωση και θα τη βάλουν στο δρόμο της ε, ενταξιακής διαδικασίας, κάτι που αξίζουν οι πολίτες της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάνοκ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Μακεδία, Μακεδονία είναι μια ευάλωτη χώρα. Με την κρίση της μετανάστευσης να έχει βασική χώρα διέλευσης αυτήν ακριβώς την περιοχή, μέσω της Ελλάδα, για πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων που μετακινούνται τις τελευταίες, τους τελευταίους μήνες. Η αστάθεια της χώρας και η άδικη μεταχείριση τη χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια που δεν τη επέτρεψαν να προχωρήσει σε διαπραγματεύσει για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια μεγάλη πρόκληση Ελπίζουμε ότι οι εκλογέ που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2016 και μια νέα κυβέρνηση θα επιτρέψουν να σταθεροποιηθεί αυτή η μικρή χώρα την οποία έχω επισκεφθεί επανελειμμένω. Η Μακεδονία έχει πολλά πολιτικά προβλήματα, όπω τα περισσότερα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή την σωστή ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, την υψηλή διαφθορά, την διαφθορά του δικαστικού συστήματο και την έλλειψη ελευθεροτυπία και ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Η έκθεση Βάγκελ καταγράφει πολύ σωστά τα αρνητικά σημεία και τα επιτάγματα τη Μακεδονία και η ομάδα μου, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, είναι πραγματικοί φίλοι τη Μακεδονία και θέλουμε να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας αυτής. Ευχαριστώ. Σακουφαρά. Κυρία Σακοράφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάγκλη, στις αρχές του χρόνου συζητήσαμε την ετήσια έκθεση πρόοδου της ΦΥΡΟ και είχα τονίσει τότε ότι η πολιτική της επιβράβευσης όλων αυτών των αρνητικών που συνθέτουν την κατάσταση της χώρας από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να μην χαθεί το momentum, όπως υποστηρίζεται, μόνο ανασταλτικά θα μπορούσε να λειτουργήσει την πρόοδό της. Του μήνε που μεσολάβησαν υπήρξε σαφή οπισθοδρόμηση και έλλειμμα σε κέριου μίσου, όπω είναι το κράτο δικαίου, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, η ελευθερία τη έκφραση, τη κατάσταση και τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη κ.ο.κ. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να μην πληρούν τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Στην παρούσα έκθεση, παρά το ότι ουσιαστικά δεν είστε σε θέση να επαναλάβετε τη θετική σύσταση για έναρξη των διαπραγματεύσεων για του λόγου που αναφέρθηκαν, στην ουσία επιβραβεύεται την μερική πρόοδο στην πολιτική συμφωνία Ιουνίου-Ιουλίου, θέτοντα σαν προπόθεση για την σύσταση έναρξη των διαπραγματεύσεων όχι τα εν πολιτικά κριτήρια αιρεσιμότητα και τα βασικά προεπαιτούμενα όπω οφείλεται, αλλά την υλοποίηση τη πολιτική συμφωνία και των επιγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων, περιορίζοντά την σε ένα και μόνο στόχο που είναι αυτό τη διαξαγωγή των εκλογών. Κλείνοντα, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά, ώστε να γίνει κατανοητό από όλου, πω το ονοματολογικό δεν αποτελεί γενικά και αφηρημένα ένα διμερέ ζήτημα μεταξύ Ελλάδα και Φύρομ, όπω θέλουν ορισμένοι εδώ μέσα να παρουσιάζουν και όπω αποτυπώνεται για παράδειγμα στην ατολική σκέψη ή τη έκθεση, αλλά ένα διεθνέ ανοιχτό ζήτημα που ο μόνο δρόμο για την επίλυσή του είναι η συνέχιση διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ η επίλυση του ΔΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελούν, όσο και ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να το ξεχνούν, ουσιώδε στοιχείο τη διαφρυσιανική διαδικασίας και της διαδικασίας σταθεροποίηση και σύνδεσης και άπτεται θεμάτων περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητα, Με πράξεις και δηλώσει που επηρεάζουν αρνητικά τι σχέσει καλή γειτονία συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών επίλυσης του ονοματολογικού, το μόνο που καταφέρνουν είναι να υπονομεύουν τι σχέσει καλή γειτονία και την περιφερειακή συνεργασία, τα οποία είναι και τα βασικά προαπαιτούμενα τη ενταξιακής διαδικασία. Η επιβράβευση τέτοιων πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων και με τη χρήση του όρου Macedonian, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση υποδαβλίζει και την εθνικιστική φρενίτιδα που επικρατεί στη χώρα, αλλά και συντηρεί τη δυσμενή κατάσταση τη χώρα που περιγράφει το ψήφισμα. Επιτρέπει στην πολιτική ελίτ τη ΦΥΡΟΜ να καλλιεργεί το έλλειμμα ανάπτυξη απαραίτητη πολιτική κουλτούρα, του σεβασμού των κανόνων δικαίων και του συμβασμού, να επενδύει στην επινόηση τη παράδοση, να αντιστρατεύεται τι θεμελιώδει αρχέ τη διεθνού ένωμη τάξη και να αγνοεί την έλλειψη πρόοδου στι καλή γειτονία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα με αυτέ τι πολιτικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, thank Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Μην ξεπερνάτε το δίλεπτο. Ο κύριος Σαφχόιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Με τόσο έλεγχο και στο Θαλής, στο τρένο. Έχω Τρεις παρατηρήσεις για την έκθεση αυτή. Προφανώς επί της ουσίας δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε με τη διεύρυνση. Δεν θα ξανασχολιάσω το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε προφανώς κατά οποιασδήποτε τρέχουσα πολιτική υπέρ τη διεύρυνσης από την ομάδα μα, Έχω όμω και κάποιε επιμερου, επιμερούς να κάνω. Στο σημείο 9, ο νόμο κατά της προπαγάνδας ε, στο εξωτερικό. ο νόμο αυτό κατά της προπαγάνδας, τη ξένης προπαγάνδας, σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών και όλοι οι νόμοι που έχουν εγκριθεί ε, μετέπειτα, έχουν αντιγραφεί ε, σαν φωτοτυπίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχύει και για τη Ρωσία και για την Ινδία αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκίνησαν αυτού του νόμου περί ξένη προπαγάνδα. Επίση θέλω να σταθώ και στο σημείο 13, όπου μιλάμε για τους Ρωμά, τις γυναίκε και τους ΛΟΑΔ. Εδώ να θυμίσω και το δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα, την θρησκευτική ταυτότητα και την χριστιανική μας ε, ταυτότητα. Είναι θεμελιώδε δικαίωμα και αυτό. Ε, το σημείο 19 επίσης πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι η Μακεδονία είναι μια χώρα με δυσχέρειες. Προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσει τις ζωές μεταναστών και αυτό προκαλεί τριγμού. Ε, αυτά τα σημεία στα οποία ήθελα να σταθώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχουμε έξι ακόμη ομιλητές στο κατάλογο και τον ολοκληρώνουμε. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εφόσον ο στρατηγικός αντικειμενικός σκοπός των Σκοπίων είναι να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, θεωρώ δεδομένο ότι η κυβέρνηση της χώρας αυτής θα κάνει ό,τι απαιτείται ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει όλες αυτές τις ισχέρειες που υπάρχουν και, όλες αυτά, όλα αυτά τα μειονεκτήματα που υπάρχουν μέχρι στιγμής τα οποία ανέφερε και ο εισηγητής και οι υπόλοιποι. Εκείνο το οποίο διαρωτώ με είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση των Σκοπίων ούτως ώστε να καθιερώσει να δημιουργήσει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα που όπως ξέρετε είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που προβλέπουν και τα κριτήρια της Κοπενχάγης για να γίνει αποδεκτή μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορέσει να αλλάξει η πολιτική και να πάψει να προκαλεί πλέον την Ελλάδα διότι πέραν της χρήσης του ονόματος Μακεδονία το οποίο όλοι γνωρίζετε και το έχουμε κατ' επανάληψη επισημάνει ότι εκφράζει επεκτατικές βλέψεις της χώρας αυτής κατά της Ελλάδος υπάρχουν και ανανεούμενες και συνεχείς προκλήσεις της χώρας αυτής κατά της Ελλάδος. Ε, δίνουν, φτιάχνουν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, δίνουν τα ονόματά τους σε οδούς και πλατείες. Πρόσφατα έφτιαξαν ένα αρχαιολογικό μουσείο και το ονόμασαν Μουσείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτω από άλλες προϋποθέσεις, εμείς ως γείτονες και ως Έλληνες θα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχείς που θαυμάζουν και αποδίδουν τις τιμές αυτές στο μεγάλο Έλληνα στρατηλάτη. Όμως πρακτικά και επί της ουσίας αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Και πώς είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός, δεχόμενος αυτές τις προκλήσεις, να επιτρέψει στην κυβέρνησή του να υπογράψει την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε ουτοπιστές για να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν αλλάξει πρακτική και τακτική, εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε στην επιβράβευση αυτής της παρανομίας. Σας ευχαριστώ. κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαγκούτκο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, ε, τον κύριο Βάγκλ, για την εκπόνηση της έκθεσης που θα συζητήσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Η Μακεδονία είσαι αρκετά ταραχώδης ε, μήνες και μετά τη συμφωνία της Οχρήτας του 2001 σίγουρα είναι η πιο τρικυμιώδης εποχή για τη χώρα αυτή. Θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Βάγκλ, ε, τον κύριο Κούκαν και τον κύριο Χόιτ ε, μαζί με τον Επίτροπο Χάν γιατί κατέβαλαν τεράστιες διπλωματικές προσπάθειες τους τελευταίους μήνες προκειμένου να καταλήξουν στη Νέα Συμφωνία Ιουνίου-Ιουλίου για να επανέλθουμε στην πολιτική σταθερότητα στη Μακεδονία και περιμένουμε τις πρόορες εκλογές του Απριλίου που ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της χώρας και στην επαναφορά της στη δημοκρατική κουλτούρα μια και έχει βλέψεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή, ε, στην, ε, έχει βλέψεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό θα ήταν να τη στηρίξουμε σε αυτό το δρόμο. Ακούσαμε τις απόψεις του κυρίου Πέτερλε ε, από την κυρία Πετήρ. Ο κύριος Πέτερλε βρίσκεται σε περιοδία στα Σκόπια Ακούσαμε λοιπόν ποια είναι η γνώμη του ΕΛΚ. Νομίζω ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ε, γιατί πολύ καθυστέρησαν τη Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να αλλάξει επιτέλους θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να απελευθερώσει το δρόμο για να μπορέσει η Μακεδονία να ξεκινήσει τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις και φυσικά εναπόκειται στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση Μακεδονίας να εκπληρώσουν τις υψηλές δημοκρατικές προδιαγραφές και να συνεχίσουν να έχουν ποιοτικέ επαφέ με τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 500.000 άνθρωποι πέρασαν του τελευταίου μήνε από την χώρα αυτή και παρόλα αυτά κατάφερε ω χώρα διέλευση να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο προσφυγικό Νομίζω ότι χρήζει τη στην υποστήριξή μας στο δρόμο της προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσκι που εκπροσωπεί τον σκιώδη συγγητή κύριο Χόουιτ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε την συνεργασία προ τη στήριξη με τον, ε, κύριο, με τον βασικό συγκεκριτή. Ο κύριος Χόουιτ έχει πολύ καλή συνεργασία μαζί του και ανυπομονή στην επόμενη, για την επόμενη επίσκεψη στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στις αρχές του Ιανουαρίου 2016. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ανησυχεί ιδιαίτερα με την ε, υποβάθμιση των πραγματών στην ε, κατάσταση αυτή ε, και αυτό ε, πολύ σωστά εντοπίστηκε και ως προς το σκάνδαλο των ε, μαζικών τηλεφωνικών αποκλειπών. Ο κύριος Χάουιτ είναι ε, πολύ ικανοποιημένο με το γεγονός ότι τουλάχιστον επετέφθη συμφωνία και συμμετείχαν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Το θέμα είναι όμως πώς θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και να μην επιτρέψουμε στην, σε διάφορα συμφέροντα να παρεμποδίσουν την επιτυχία της συμφωνίας. Ως προς την έκθεση του κυρίου Βάγκλη θα υποβάλουμε μια σειρά από τροπολογίες, θα τις συζητήσουμε και κατηδίαν και με τον κύριο Βάγκλη και ήδη Ξέρουμε ότι ο κύριος Χάν έχει ε, ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων για την διεύρυνση ήδη φέτος, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να δούμε ότι έχουν διοργανωθεί ανεξάρτητα και δικαίως οι εκλογές. Η κατάσταση στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει γίνει θετικότερη. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και με αυτή τη χώρα πολύ αυστηροί με τα κριτήρια ε, διεύρυνσης και ένταξης όπως έχουμε υπάρξει καθένα. Ευχαριστούμε επειδή μας πήγαινε να λέει το χρόνο σε ένα λεπτό για τον καθένα. Ο κύριος Όλτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγκλη για το κείμενο της έκθεσης που είναι άριστο το ψήφισμα αυτό για τη Μακεδονία η Μακεδονία που είναι ήδη υποψήφια χώρα εδώ και 10 χρόνια και θεωρείται ως μία από τις πιο προηγμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι λοιπόν για μένα κρίμα να παρεμποδίσουμε την ένταξη της χώρας αυτής μόνο και μόνο λόγω της ονομασίας της. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η Μακεδονία θα πρέπει να βρουν ε, μια λύση σε αυτό το διέξοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στηρίζει τη Μακεδονία και θα τη στηρίξει σε όλη την πορεία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένταξη και θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ότι μισό εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν από την επικράτειά της τους τελευταίους μήνες και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χώρα αυτή για την σταθερότητα στην όλη περιοχή. Οι πρόσφυγες περνούν από ένα κράτος μέλος πρώτα, μετά από την Μακεδονία, μετά από ένα άλλο κράτος μέλος. Πρέπει λοιπόν και η Frontex να στηρίξει τη Μακεδονία και να υπάρξει οικονομική βοήθεια. Ε, η πολιτική κρίση της Μακεδονίας φέτος βέβαια ήταν πολύ σοβαρή, αλλά χάρη και στη συμμετοχή των δικών μας ε, συναδέλφων, των Ευρωβουλευτών, ε, βρέθηκε μια λύση για την κρίση αυτή. Υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη ότι η κατάσταση θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί εντωμεταξύ, παρόλο που αναμένουμε ακόμη εντατικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, στον τομέα των μεσονομικής ενημέρωσης, στην δημοσιαδίκηση και χρειάζεται και μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς από την δική μα πλευρά. Ο κύριο Κοβάτσεφ για ένα λεπτό. Θα είμαι λακωνικός ε, κύριε Πρόεδρε. Δύο σημεία. Καταρχήν για όλες τις γειτονικέ χώρες αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία ε, της Μακεδονίας, ιδιαίτερα με τις προκλήσεις ε, που μας δημιουργεί το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό. Θέλουμε ελευθεροτυπία, πάταξη των διακρίσεων, πάταξη της διαφθοράς, καταπολέμηση της διαφθοράς και επαναφορά του κράτους δικαίου. Αλλά να σταματήσει η, επιλεκτική ερμηνεία των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σταματήσει η παραπλάνηση των ιστορικών γεγονότων στα σχολικά βιβλία. Γιατί ο εθνικός χαρακτήρας ε, της περιοχής της Μακεδονίας είναι πολυεθνικός. Η μακεδονική σαλάτα τι σημαίνει. Σημαίνει μια σαλάτα με πάρα πολλά συστατικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Μακεδονίας. Έχουμε ιστορική παρουσία της βουλγαρικής κοινότητας ε, που από το, ε, από το 1944 παρουσιάζονται ως Μακεδόνες. Ευχαριστώ κύριε Σανδρουλάκης. Για το ονοματολογικό βλέπω ότι υπάρχει αναφορά με την οποία καλείται η εκπρόσωπος να εμπλακεί περισσότερο στη διαδικασία επίλυσης του καθώς και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς της. Παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικό να έχει ενημέρωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι καλοδεχούμενη, οφείλω να υπογραμμίσω ότι το μόνο κατάλληλο πλαίσιο για την επίλυση του νοματολογικού είναι αυτό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο φόβο μου είναι ότι οποιαδήποτε εμπλοκή τη ύπατη εκπροσώπου ενδεχομένως να στείλει λάθο μηνύματα στη ΦΥΡΟΜ να δυσχεράνει προσπάθειε επίλυση του ομαδολογικού ζητήματο παρά τι οποίε καλέ προσπάθειε. Επιπροσθέτω, πρέπει να αναφερθούμε και στο ζήτημα τη μη αναφορά στι σχέσει καλή γειτονία, η σημασία των οποίων είναι φυσικά αδίρετη... και, περι... και περιλαμβάνει το θέμα του ομαδολογικού. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα των κριτηρίων τη Κοπεχάγη και των λοιπόν προαπαιτουμένων, οφείλω να υπογραμμίσω ότι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι απαραίτητη η εκπλήρωση τους και δεν νοείται σχετική αίρεση. Με αυτά σχετίζονται ζητήματα όπως η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, της δικαιοσύνης, η ελευθερία έκφρασης και προφανώς η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν που μιλάει στο όνομα του κυρίου Κούκαν. Εκπροσωπεί τον εαυτό του δηλαδή ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση Βάγκλ και να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του, αλλά και για τη συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία διευκόλυνσης ε, του ΕΛΚ. Ελπίζω οι Μακεδόνες πολιτικοί να δείξουν το θάρρος και την πολιτική βούληση να ξεπεράσουν αυτή την κρίση. Θα είναι σημαντικό για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να επαναφέρουμε τη χώρα την ενταξιακή διαδικασία, κάτι που θα απαιτήσει προσπάθειες και από δική μας πλευράς, αλλά κυρίως ε, την ε, επικοδομητική ε, συμπεριφορά και δέσμευση όλων των πολιτικών παραγόντων της χώρας. Συμμετείχα στη διευκόλυνση της σύναψης της συμφωνίας, γι' αυτό και απευθύνω έκκληση ε, για την εφαρμογή της Συμφωνίας 2 ε, Ιουνίου 15 Ιουλίου γιατί είναι ο δικός χάρτης για την επαναφορά της χώρας στη σταθερότητα αλλά και την ε, εκ νέου επαναφορά στην ενταξιακή διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριος Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βάγγελ για αυτήν την έκθεση λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις της Κομισιόν. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα. Από την έκθεση πρόοδου της φετινής χρονιάς προκύπτει ότι τα προβλήματα διαφοράς, η καταπάτηση των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, της ελευθερίας έκφρασης αποτελούν αντικείμενο διατυπωμένων συστάσεων. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή η Μακεδονία πρέπει να υποστηρίξει το δικαίωμα να μιλά κανείς τη μητρική του γλώσσα. Πρέπει να καταλάβει η άρχουσα ελίτ των Σκοπίων ότι υπάρχουν κανόνες αν θέλουν να ενταχθούν προοπτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα με τι διαπραγματεύσεις των Σκοπίων δεν είναι η ονομασία, είναι το έλλειμμα δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό άλλωστε είπε και η Επιτροπή, ότι δεν σέβεται τα κριτήρια της Κοπεχάγης, δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν σέβεται τα θέματα της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει θεωρία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν υπάρχει διαφθορά. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα Σκόπια. Όσον αφορά την ονομασία, σε διμερέ επίπεδο βεβαίω ο καθένα, αφού η χώρα του έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, α κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι διμερέ, το πρόβλημα είναι διεθνέ και πρέπει να επιληθεί μέσα στα πλαίσια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι και η θέση τη Επιτροπή. Θα σας, θέλω να σα κάνω μια παρατήρηση ως συμβολή στη δικιά μου παρέμβαση στη συζήτηση. Έχει δίκιο ο κ. Κοβάσεβιτ όταν λέει ότι εκεί είναι μια μακεδονική σαλάτα. Γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δικαιώσουμε την πολιτική του Τίτο του 1944 που ήθελε να δημιουργήσει εκεί ένα κράτος. Όταν μιλάνε, το είδα στη Βουλγαρία αυτό, του λέει ο Βούλγαρος συνάδελφος γιατί δεν μιλάς τη μητρική σου γλώσσα αλλά μιλάς αγγλικά. Και η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της γλώσσας αν μιλήσουν θα καταλάβουν οι Βούλγαροι συνάδελφοί μου. Το ίδιο πράγμα έγινε με την Εκκλησία και το ίδιο πράγμα έγινε με την ονομασία για, την, για το Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι γεωγραφικό προσδιορισμό, δεν μπορεί να καπηλεύεται και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να δικαιώσουμε την πολιτική του τίτλου ενό αυταρχικού καθεστώτο εκείνη τη εποχή. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για σύντομα παρακαλώ σχόλια. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αντιμετωπίζει την σοβαρότερη πολιτική κρίση της εδώ και χρόνια. Η πολιτική συμφωνία που υπεγράφει από τους ηγέτες έχει τεθεί σε ισχύ και αυτό διευκολύνθηκε από τον Επίτροπο Χάν και τους ε, Ευρωβουλευτές Κούκαν και Βάιγκλ, τους οποίους εκτιμούμε πολύ. Τον Ιούνιο η Κομισιόν παρουσίασε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων επίγουσας ε, σημασίας κυρίως στο κράτος δικαίου. Έχει ξεκινήσει το έργο, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Φέτος, υπό το φως ε, της προόδου που επετέφθη σε αυτήν την ε, συμφωνία, η Κομισιόν ε, προτίθεται να ανοίξει τις ε, να, να προβεί σε σύσταση για άνοιγμα των διαπραγματεύσεων ε, για ένταξη στην Ένωση. Αυτό όμως υπό τον ε, όρο της εφαρμογής συμφωνίας του Ιουνίου και των μεταρρυθμίσεων. Η Κομισιόν θα περιμένει έως τις εκλογές της επόμενης χρονιάς. Στο μεσοδιάστημα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της χώρας και καλούμε τους ηγέτες να ενεργήσουν ε, υπέρ του συμφέροντος της χώρας και των πολιτών της. Κύριε Βάιγκλ, παρακαλώ για τις ε, παρατηρήσεις σας για να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν σε αυτή τη συζήτηση και συμμετείχαν. Μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περιοχή της Ευρώπης. Από καιρού εις καιρόν αυτό προκαλεί προβλήματα και στην υπόλοιπη Ήπειρο. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι η Μακεδονία και οι γειτονικέ της χώρες να γίνουν ένας παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας για την Ευρώπη. Μου φαίνεται λοιπόν σημαντικό όλες αυτές οι χώρες να μπορούν να συνεργαστούν, να οικοδομήσουν από κοινού μαζί μας την Ενωμένη Ευρώπη. Έχουν γίνει πολλές σύνοδοι στο Συμβούλιο και έχουν ακουστεί και πολλά θετικά σχόλια, πολλές καταφατικές υποσχέσεις αλλά και πολλά επικριτικά σχόλια για τη Μακεδονία. Παρακολουθώ ιδιαίτερη προσοχή όλες τις προτάσεις για το πώς θα πρέπει να ε, συμπληρωθεί η έκθεση αυτή και θα συνεργαστώ με όλους όσοι επιθυμούν να βελτιωθεί για να έχουμε το καλύτερο δυνατό ψήφισμα. Θα ήθελα απλώς να κάνω μια σύντομη παρατήρηση για τα διάφορα γαστρονομικά που ακούστηκαν, δηλαδή πέραν του μεγάλου πλούτου της όλης γεωγραφικής ε, περιοχής, έχει μια ποικιλία από σαλάτες η όλη περιοχή να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ελληνική, τη μακεδονική, την ε, λεγόμενη σέψκα και επίσης και μια σειρά από καφέδες, τον ελληνικό, το σερβικό Όλος αυτός λοιπόν ο πολιτιστικός πλούτος της περιοχής, ακόμη και από γαστριμαργική σκοπιά, είναι πραγματικά προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Θα ήθελα τώρα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών έχει οριστεί για τις 14 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, που προβλέπει την έκθεση προόδου του 2015 για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που επίσης αντιμετωπίζει δύσκολες προκλήσεις φέτος, αλλά έχει και θετικές εξελίξεις, όπως η πρόσφατη πρόσκληση του ΝΑΤΟ για ένταξη, αλλά είχαμε και αρνητικέ εξελίξει, ε, σημαντικέ εντάσει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάτι που οδήγησε σε μια πολιτική αστάθεια, καθώ και το μποϊκοτάρισμα τμήματο τη αντιπολίτευση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση και προς την κυβέρνηση και προς το δημοκρατικό μέτωπο να ε, συνεχίσουν ε, τον επικοδομητικό διάλογο και μια καρποφόρα συνεργασία στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή διαδικασία, το Μαυροβούνιο εξακολουθεί να σημειώνει σταθερή πρόοδο και μάλιστα είναι η πιο προηγμένη χώρα σε ό,τι αφορά το ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, έχει και σημαντικές ευθύνες ε, στην περιφέρεια σε ό,τι αφορά την ε, γενικότερη ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, βέβαια υπάρχουν ακόμη κάποιες προκλήξεις στην ενταξιακή διαδικασία. Πόλωση του πολιτικού κλίματος, πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης και υπερβολική πολιτική ε, επιρροή στη δικαστική εξουσία, ε, πρόβλημα στην ελευθεροτυπία, διαφθορά και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τσάρλς Τάρνοκ είναι ο εισηγητής που θα αναλύει τα τα ισχυρά και τα δύναμα σημεία του Μαυροβουνίου και την έκθεση πρόεδρε του 2015. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου γιατί εξακολουθώ να είμαι ε, ο εισηγητής για το Μαυροβουνίο που είναι σχετικά ε, εύκολη υπόθεση σε σχέση με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια γιατί συνεχίζει την σταθερή πορεία ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου σε υποψήφια χώρα για την ένταξη. Και μάλιστα πρωτοστατεί σε σχέση με τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Έχει ανοίξει 20 διαπραγματευτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων 23 και 24. Βέβαια τα θέματα διαφθοράς υψηλού επίπεδου και οργανωμένου εγκλήματος εξακολουθούν να δημιουργούν τεράστιε προκλήσει, αλλά σε όλου σχεδόν του τομεί, έχουμε διαπιστώσει πρόοδο στην ανάπτυξη των ε, θεσμικών οργάνων, στη μεταρρύθμιση τη δικαστική εξουσία, αλλά και στην ε, εφαρμογή των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ένα στενές ευρώ που χρησιμοποιείται ως de facto νόμισμα στο Μαυροβούνιο βοήθησε τη χώρα αυτή και διευκόλυνε τον τουρισμό της. Και μάλιστα ενισχύθηκε ο τουρισμός επειδή άλλοι τουριστικοί προορισμοί όπως η Τουρκία, η Τινησία και η Αίγυπτος εξαιτίας των τρομοκρατικών απειλών ήταν ε, μια μείωση του τουρισμού τους. Εποφελήθηκε αυτό, από αυτό την κατάσταση στο Μοντενέγρο που είχε μια πολύ καλή τουριστική εποχή. Βέβαια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία ε, δεδομένης και της κρίσης στην περιοχή. Και το γεγονός ότι κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκότερα φέτος στο Κοινοβούλιο δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες. Γι' αυτό και θα ήθελα να απευθύνω και εγώ έκκληση, όπως και ο Επίτροπος και άλλοι, σε όλα τα πολιτικά κόμματα του Μοντενέγκρο να συμμετέχουν σε δημοκρατική συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου και να μην μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στους δρόμους. Και μάλιστα η πρόσκληση του ΝΑΤΟ της περασμένης εβδομάδας προς το Μοντενέγκρο για να ενταχθεί στη Διαδηλατική Συμμαχία είναι σημαντικό βήμα ε, και σημαντική ευκαιρία να ευθυγραμμίσει ε, η χώρα αυτή την αμυντική πολιτική της με τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Επίσης ε, συμμετέχει στις κυρώσεις της Ευρώπης προς τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας και την κατοχή της κοιλάδας του Ντουναβιντόμπας. Συνεχίζουμε του Ντονέσκ, συγγνώμη. Ε, συνεχίζονται οι ε, διαδικασίες αυτές ε, ένταξης ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν ε, μεγάλα κενά σε ό,τι αφορά τους στόχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μαυροβούνιο έχει ένα μικρό αλλά σημαντικό πρόβλημα ριζοσπαστικοποίησης και ε, πολλοί κάτοικοι του ε, έχουν αναφερθεί ότι είναι τζιχαντιστές και πολεμούν στο πλευρό του Ισλαμικού Κράτου. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση γνωρίζει το θέμα και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ την κατάσταση. Περιμένουμε ανυπομονησία τα σχόλια των συναδέλφων σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση πρόοδου. Ε, εδώ και 6 χρόνια είμαι ο εισηγητή ε, για το Μαυροβούνιο και πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στη συνένεση και να... σε ένα θετικό ψήφισμα για την πρόοδο του Μαυροβουνίου για την ε, συνταξιακές διαπραγματεύσεις φέτος. Είναι μικρή χώρα και μεγάλη επιτυχία της μετά την ανάκτηση ανεξαρτησίας. Και είναι ο καλός μαθητής στα Δυτικά Βαλκάνια σε ό,τι αφορά την ανταξιακή διαδικασία. Βέβαια έχει τεράστια προβλήματα τους τελευταίους μήνες εξαιτία τη τεράστια προσφυγική προσφυγικής κρίσης. Βέβαια δεν είναι άμεσα χώρα διέλευσης, αλλά έμεσα έχει επηρεαστεί από το προσφυγικό και από τις ταραχές ε, τις πολιτικές που κυριάξαν στη χώρα. Πάρος, εγώ είμαι θερμός υπέρμαχος του Μαυροβουνίου και ευελπιστώ ότι κάποια μέρα θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συντομότερο δυνατό. Περιμένω τα σχόλια των ε, συναδέλφων και φυσικά και τις ενδιαφέρουσες τροπολογίες τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καν εκ μέρους της κυρίας Ντότς, πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του, Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου με το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή, η οποία έρχεται σε σημαντική στιγμή λόγω και της ε, θερμής πολιτικής κατάστασης στο Μαυροβούνιο. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το διάλογο τους στο Κοινοβούλιο. Επίσης, οι ειρηνικές ενέργειες αποτελούν συστατικό μια ε, μιας δημοκρατίας. Οι πράξεις βίας στις πρόσφατες διαδηλώσεις θα πρέπει να διερευνηθούν. Θα γίνουν προώρες εκλογές την επόμενη χρονιά στο Μαυροβούνιο και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα θα είναι η εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου προκειμένου να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές διαδικασίες. Οι μαυροβουνιοί πολιτικοί θα πρέπει να συνεργαστούν για το στόχο αυτό και να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν με άψογο τρόπο το νέο σύστημα είναι πολύ απαιτητικό και είναι σημαντικό να ξεκινήσει η δουλειά από τώρα ώστε το σύστημα αυτό να είναι αρκετά ανθεκτικό την ημέρα των εκλογών. Τρεις, τρία χρόνια μετά την έκθεση που είχε εκδοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει δοθεί συνέχεια. Ζήτημα διαφθορά. Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά δεν έχουν υπάρξει παρά μόνο λίγες για υψηλά ματούχους. Και τέλος, ανησυχώ για το γεγονός ότι το Pride της ΛΟΑΤ κοινότητας έχει απαγορευτεί τη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. You it's time for, uh, rapporteurs, Τώρα τους και ό,τι Ο κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τάνοκ για την έκθεσή του. Είναι από τα πιο ισορροπημένα ψηφίσματα που έχουμε δει για το Μοντενέγρο. Και συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ ότι το Μοντενέγρο, το Μαυροβούνιο είναι ο καλός μαθητής των Δυτικών Βαλκανίων. Κάτι που δεν θα πρέπει να προκαλέσει τη ζηλετοφθόνο των γειτονικών χωρών, αλλά ίσα ίσα να του δώσει κίνητρα και να δημιουργήσουν μια άμυλα με το Μαυροβούνιο. Φυσικά η νέα εκλογική νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί και όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν και πάλι μέρος σε ένα επικοδομητικό πολιτικό διάλογο προκειμένου να συντρέξουν και τα οικονομικά κριτήρια και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας γιατί και η ανεργία είναι υψηλή και το δημόσιο χρέος. Επίσης, ε, χρειάζεται και μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας αλλά και μεταρρύθμιση στη δικαστική εξουσία και στη δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που θεωρητικά υπάρχουν. Βέβαια, η πολιτικοποίηση σε μια χώρα με μόνο 600.000 κατοίκους είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει ε, να συνεχιστεί η προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να αποδειχθούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Βέβαια, έχουμε προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιορισμένη ελευθερία έκφρασης και άσκηση βίας κατά των δημοσιογράφων. Ε, η μυσαλλοδοξία επίσης θα πρέπει να περνά παρατήρητη ή ατιμόρυτη. Χαίρομαι που το Μοντενέγρο ευθυγραμμίστηκε με την ευρωπαϊκή πολιτική στην κρίση της Ουκρανίας και στην πολιτική κατά του Ισλαμικού κράτους. Χαίρομαι για την πρόσκληση του ΝΑΤΟ να προσχωρήσει το Μαυροβούνιο, αλλά είδαμε ότι η Ρωσία και πάλι επιχείρησε και στην περίπτωση του Μαυροβουνίου να κάνει αρνητικά σχόλια για αποφάσεις που κανονικά είναι αποφάσεις κυρίαρχου κράτους ε, να προσχωρήσει σε μια πολιτική ή στρατιωτική συμμαχία. Είναι απαράδεκτα αυτά τα αρνητικά σχόλια που έκανε η Μόσχα. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Τάνοκ για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσίασε είναι μια πολύ καλή βάση και είμαι σίγουρος ότι θα επαναλάβουμε την καλή συνεργασία που είχαμε την προηγούμενη χρονιά το Μαυροβούνιο έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο. Φέτο ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει σε τέσσερα καινούργια κεφάλαια, άνοιξαν φτάνοντα στο συνολικό αριθμό των 20, εκ των οποίων τα δύο έχουν προσωρινά κλείσει. Η πρόοδο που έχει επιτευχθεί μπορεί να διαφανεί και στην έκθεση πρόοδου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω, παρά την πρόοδο, πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα στον τομέα τη καταπολέμηση διαφθορά, του οργανωμένου εγκλήματο και του πελατειακού κράτους. Δυσάρρωστο γεγονό αποτελεί και η απόφαση κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης να απέχουν από τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Ο πολιτικός διάλογος είναι αναγκαίος και πρέπει να γίνεται εντός του Κοινοβουλίου. Είναι αναγκαίο επίσης να διασφαλιστεί η διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών βάσει του νέου εκλογικού νόμου που δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονική ταυτοποίηση των εκλογέων. Δυστυχώ παρά τα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερα την αύξηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα, η ανεργία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειε για την εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και των περιστατικών βία εναντίον των ΛΟΑΤ. Στα θετικά τέλο, πρέπει να προσμετρηθεί και το γεγονό ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί ίσω τη μόνη υποψήφια προσένταξη χώρα της οποίας η εξωτερική πολιτική συμβαδίζει σχεδόν στο 100% με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου στηρίζει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Rados. Ράντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να επενέσω τον κύριο Τάνοκ για την πολύ καλή του έκθεση και τα κλασικά ζητήματα όπως τα καλύπτει, όπως ε, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, τη διαφθορά, την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος, την κοινωνία των πολιτών και την ελευθερία του μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα αντιμετωπίζει με πολύ ισόρροπο τρόπο. Να τονίσω δύο πολύ σημαντικά για μας πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πρόσκληση προς το Μαυροβούνιο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ έχοντας υπόψη ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ωφέλιμη για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και το θέμα των εκλογών. Ε, νέες εκλογές με υψηλές δημοκρατικές προδιαγραφές που θα είναι ευεργετικές για τις μακροχρόνιες, σταθερές και θετικές σχέσεις μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης. Ίσως του χρόνου να υπάρξουν τέτοιες εκλογές στο Μαυροβούνιο. Thank you, uh, Χατζηγεωργίου. Καλημέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τάνοχ για την εργασία του για έκτη συνεχή χρονιά. Φαίνεται ότι η χώρα για την οποία συζητάμε είναι σε καλή πορεία προς την ένταξη. Υπάρχουν προβλήματα δημοκρατίας στη χώρα, όπως μάλλον υπάρχουν και σε πολλές χώρες που είναι ήδη ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει να κάνει με τις σχέσεις αντιπολίτευσης-συμπολίτευσης ή με τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης, είτε του δικαιικού συστήματος. θέλω μόνο να βάλω μια ένσταση και να την δικαιολογήσω. Η πρόταση στην έκθεση που καλεί την χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι είναι μια κακή προσέγγιση. Έστω και αν αυτό είναι μια συνήθις διαδικασία, δηλαδή στο Κοινοβούλιο το βλέπουμε σαν αυτό να είναι φυσικό επακόλουθο της ένταξης οποιοδήποτε κράτους. Ο λόγος που είπα να το εξηγήσω είναι για να πω το εξή. Εμείς δεν είμαστε υπέρ οποιοδήποτε συμφώνου της Βαρσοβίας, για παράδειγμα. Είμαστε ενάντια σε στρατιωτικές συμμαχίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν είναι υποβοηθητικές για την ειρήνη. Η τάση επέκτασης του ΝΑΤΟ προς την κατεύθυνση της Ρωσίας, όσο και αν κάποιοι την κρίνουν δικαιολογημένη και δεν μπαίνω σε αυτό, ουσιαστικά προκαλεί εντάσεις, πολέμους και αίμα και νομίζω πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό. Γι' αυτό η έκκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ θεωρούμε ότι είναι ε, Ευχαριστώ. Ε, thank you, Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου των Πρασίνων να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τάνοκ για μια πολύ καλή έκθεση που ε, απαντά σε δύο πράγματα. Ε, τις θετικές προοπτικές του Μαυροβουνίου που έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από άλλες χώρες όσον αφορά την ενταξιακή της πορεία και εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι είστε επικριτικός στους, ε, στα θέματα στα οποία πρέπει να γίνουν πράγματα. Διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, ε, ελευθεροτυπία, η κατάσταση στην κοινωνία των ε, πολιτών. Υπάρχουν ε, κάποια σημεία στα οποία θα θέλαμε να ενισχυθεί όμως η έκθεση. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί είναι και αυτό ένα από τους ε, τομείς στους οποίους υπάρχει διαφθορά. Επίση, εκτιμώ το γεγονό ότι ζητείτε περισσότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί εμείς ως ε, βουλευτές ε, πρέπει να το υποστηρίζουμε αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που θα ήθελα να ε, προσθεθούν στην έκθεση. Για παράδειγμα, ότι η Επιτροπή Καταπολέμησης τη Διαφθοράς στο Κοινοβούλιο έχει μπλοκαριστεί λόγω της πλειοψηφίας των κυβερνητικών κομμάτων στην Επιτροπή αυτή, η οποία δεν είναι μάλιστα αναλογική ε, προς τον ε, συσχετισμό στην Ολομέλεια. Εγώ πιστεύω ότι σε μια τέτοια επιτροπή κατά πολέμησης διαφθοράς είναι πολύ σημαντικό η αντιπολίτευση να έχει λόγο. Ε, θα λάβετε όμως, δεν θα τις αναφέρω όλες, θα λάβετε πολλές, κάποιες τροπολογίες από εμάς. Επίσης, ε, χαίρομαι που ε, εντάξατε κάποια ζητήματα οικολογικής ε, φύσης γιατί το Μαυροβούνιο αναφέρει και κατοχυρώνει και στο Σύνταγμά του ότι είναι μια οικολογική χώρα. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ε, αναφέρεται το ζήτημα της ε, ε στο Ούτσιν που είναι πολύ σημαντικός χώρος αναπαραγωγής ε, πουλιών. Επίσης θα ήθελα να ε, αναφέρετε κάτι για τον σχεδιασμό μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Είχαμε κάποια ψηφίσματα και στο παρελθόν για, τον, για τα σχετικά σχέδια στον ποταμό Μόρατσα και το στρατηγικό σχεδιο, σχεδιασμό για μεγάλης κλίμακας και μικρής κλίμακας υδροελεκτρικές εγκαταστάσεις. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, υπάρχουν κάποια αποσπασματικά έργα από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό θα λάβετε και κάποιες τροπολογίες από εμά. Και κάτι τελευταίο. Για το ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι στην έκθεση προόδου σε μια έκθεση προόδου το ζήτημα του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο ρόλο. Είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι ε, το ΝΑΤΟ μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά στη χώρα. Εγώ φυσικά δεν θέλω η Μόσχα να ε, παίζει μεγάλο ρόλο ε, και δει στα Βαλκάνια. Αλλά τα χρήματα ε, Ρώσων επενδυτών βρίσκονται ήδη στη χώρα. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να εισβάλλουν οι Ρώσοι στη χώρα. Αν θέλουμε οπωσδήποτε να αναφερθούμε στο ΝΑΤΟ, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να καλούμε ε, στο να υπάρξει ένα δημοψήφισμα ε, κάτι που εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και το δημοσίευμα που θα γίνει το επόμενο διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως εγώ αυτή ε, είναι η κατεύθυνση στην οποία νομίζω ότι πρέπει να ε, κινηθούμε. Είμαστε απελπισμένοι γιατί ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα και μένουμε όλο και περισσότερο πίσω. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές τώρα. Αλλά μόνο για 1,5 λεπτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ο κύριος Αφόιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανονικά εκπροσωπώ την ομάδα μου εδώ. Θα ήθελα να πω ότι είναι πιστή η περιγραφή ε, της κατάστασης που κάνει η έκθεση Τάνοκ. Θα την καταψηφίσουμε όμω. Στο σημείο 3 μιλά για τη χαοτική πολιτική κατάσταση στη χώρα. Στο σημείο 8 μιλά για τη διαφθορά που είναι ανησυχητική. Στο σημείο 11 λέει ότι ε, δεν γίνεται σωστή δίωξη των υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος. Στο σημείο 15 μιλά για περιορισμένη ελευθεροτυπία. Παρακάτω μιλάει για τους Ρωμά, τους ΛΟΑΔ. Κάθε φορά που αναφέρουμε αυτές τις μειονότητες θα πρέπει να μιλούμε και για την πολιτιστική και πνευματική ταυτότητα γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτές τις ε, πνευματικές κοινότητες ε, και τις πολιτιστικές που θα πρέπει να τα δικαιώματά τους να γίνουν σεβαστές. Επίσης, ε, παρακάτω στο σημείο 20 αναφέρονται τα ενοχικά δικαιώματα που δεν τηρούνται. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, θα καταψηφίσουμε την έκθεση Τάνοκ. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη θέλει περισσότερο να δημιουργεί γέφυρες, αλλά όχι κατακαιρματισμό ή διχασμό της Ευρώπης στα δύο, η διχοτόμηση. Και πραγματικά δεν είμαστε εμείς σε θέση ε, ενώ υποτίθεται ότι κοπτόμαστε για την ενότητα και την ειρήνη, να θέλουμε να κόβουμε στα δύο, να διχοτομούμε την Ευρώπη ε, και να διαχωρίζουμε την Ευρώπη από τη μια και την Ρωσία από την άλλη. Και νομίζω ότι τέτοιου είδου ε, διχαστικέ πολιτικέ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα τη Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριο Πλέγκοβιτ. Ευχαριστώ κύριε Λαγκούτκο. Έχω και εγώ μερικά σχόλια για τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την πολύ σημαντική του έκθεση για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο σίγουρα ε, είναι με διαφορά η πιο προηγμένη ε, χώρα σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια στην μεταξιακή διαδικασία. 20 κεφάλαια έχει ανοίξει στις διαπραγματεύσεις και την περασμένη εβδομάδα δέχτηκε την πρόσκληση του ΝΑΤΟ για προσχώρηση στη συμμαχία αυτή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και για τη γεωστρατηγική ισορροπία της περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβω υπόψη και χαίρομαι που το ανέφερε ο κύριο Στάνοκ στην έκθεσή του. Τρίτο σημείο, η εσωτερική πολιτική κατάσταση, όπω και στι υπόλοιπε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, στη Μακεδονία, στο Κωσυφοπαίδιο και στην Αλβανία έτσι και στο Μαυροβούνιο είχαμε μαζικές διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. Πάντως είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ανταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου αμετάβλητη γιατί θα συμβάλλει στη δημοκρατική ανάπτυξη και καλό θα ήταν να στηρίξουμε τη χώρα αυτή στην ανταξιακή της πορεία. Ευχαριστώ κύριο Σπίτσουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση του κυρίου Τάνοκ. Πολύ αξιόλογο έγγραφο και πολύ ισορροπημένο. Ε, είναι εύκολο να δούμε τις ε, επιτυχίες και την πρόοδο του Μαυροβουνίου. Για παράδειγμα, 20 κεφάλαια άνοιξαν, πολύ ορατή πρόοδο. Συγχαρητήρια για την πρόσφατη πρόσκληση του ΝΑΤΟ για ένταξη. Ως ακροάτης πολιτικός χαίρομαι για τη γεωπολιτική αυτή η εξέλιξη και ότι θα έχουμε ένα νέο μέλος στο ΝΑΤΟ. Γιατί πριν 25 ε, χρόνια είχαμε εισβολή στη χώρα ε, και καλό θα ήταν να επιστρέψουμε τώρα πια στη σταθερότητα. Βέβαια, το Μαυροβούνιο έχει πολλές εκκρεμότητες να διαθετήσει. θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά να κρατήσει ανοιχτό το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και επίσης ε, θα πρέπει να επανέλθει μια ομαλή λειτουργία και πορεία στις σχέσεις ε, κυβέρνηση και αντιπολίτευση που είναι πολύ ταραγμένες αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Σουίτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την πολύ αξιόλογη έκθεσή του. Σίγουρα είναι αισθητή η πρόοδο του Μαυροβουνίου. Άνοιξαν 20 κεφάλαια για τι διαπραγματεύσει. Εκεί που μιλάτε για την πρόσκληση του ΝΑΤΟ, είναι σημαντικό αυτό το θέμα, ε, κυρίως για τις γειτονικέ χώρες ε, και για την Κροατία. Χαίρομαι που το αναφέρετε. Εγώ έχω τρία σχόλια. Αναφέρετε αναφέρετε συγκεκριμένα ονόματα σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Αναφέρετε συγκεκριμένα ονόματα. Επίσης, ε, καλό θα ήταν, μια και μιλούμε για κρωμάτες, να μιλούμε και για ένα πρόβλημα εδαφικό που δεν έχει διευθετηθεί ακόμα μεταξύ Μαυροβουνίου και Κροατίας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τα μέλη του Μαυροβουνίου που ήταν σε στρατόπεδα στη διάρκεια του πολέμου και δεν έχουν ακόμη ε, γίνει σεβαστά τα δικαιώματά τους. Είναι σημαντικό, το επισημάναμε στην προηγούμενη έκθεση, την περσινή, αλλά δεν υπήρξε καμία πρόοδος. Θα ήθελα λοιπόν να το τονίσετε αυτό, γιατί καλώς μιλάτε για την ελευθεροτυπία, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τις άλλες διακρίσεις. Υπάρχουν κάποιες ε, δεοντολογικές και ηθικές προδιαγραφές, ε, αλλά απευθύνεται έκκληση και πολύ σωστά να υπάρξει πρόοδος και στο σημείο αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερωτυπία. Ευχαριστώ κύριε Σκούκαν. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Τανόκ. για την ε, πολύ ποιότητα σε αυτή η έκθεση ως συνήθως και όταν λέω ψηλή ποιότητα εννοώ ότι αναφέρει όλα τα θετικά επιτέμματα της χώρας αλλά ταυτόχρονα και ε, το που εντοπίζονται προβλήματα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να προοδεύσει κι άλλο η χώρα. Με τον τρόπο που τα διατυπώνει, ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνουν ω τώρα και πρέπει να του θυμίζει ότι είναι από του ε, πρωταρχηγού τη διαδικασία διεύρυνση για την όλη περιοχή. Αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση, είναι υπενθύμηση ότι έχουν ευθύνε. Έχουν λάβει ευθύνε και δεν πρέπει να μα απογοητεύσουν. Νομίζω ότι πρέπει απαραίτητος να ε, αναφερθεί ότι υπάρχει 100% ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά για αυτή την έκθεση πρόοδου. Το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είναι σαφές ότι δίνουμε, θέματα, ότι δίνουμε έμφαση στα θέματα κράτους δικαίου και με μια λέξη μπορώ να πω ότι το κράτος δικαίου και ενίσχυσή του θα καθορίσει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Τώρα για το θέμα της παρέλασης ΛΟΑΔ, της Gay Pride, επειδή τέθηκε και αυτό, θα γίνει αυτή την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στην Ποντγκόριτσα, παρά την αναβολή. Σε λίγα λεπτά θα ήθελα να σας ενημερώσω και για την κατάσταση που βλέπουμε σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να επιτρέψει να υπάρξει επικοδοματικός διάλογος μεταξύ των κομμάτων αυτών. Όπως ξέρετε, ο Επίτροπος Χάν στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε διατησία. Θα πρέπει τη λύση να τη βρουν τα ίδια τα κόμματα του Μαυροβουνίου. Η πρώτη σχετική συνάντηση έγινε την 1η Δεκεμβρίου και ε, ασχολήθηκαν στις συζητήσεις με τον έλεγχο των δημοσίων κονδυλίων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με τον ε, διακομματικό διάλογο. Θα συνεχιστεί όλο το Δεκέμβριο μέχρι τις 21 η συνεργασία αυτή, όπου δεν θα ξανασυναντηθούν οι αρχικοί των πολιτικών κομμάτων με σκοπό να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον καλύτερο τρόπο να εφαρμόσουν τη συμφωνία τους. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα της απολυτεύσης εκτός από το δημοκρατικό μέτωπο συμμετείχαν στην ομάδα εργασία. Το Δημοκρατικό που είπε ότι θα συμμετάσχει στο διάλογο μόνο εφόσον σχηματιστεί μια ενδιάμεση κυβέρνηση, μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, κάτι που δεν ισχύει ως τώρα. Αλλά μπορεί να επανέλθει ως θέμα αργότερα. Δεν είναι βέβαιο τι θα συμβεί με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα λόγο πάλι στον κύριο Τάνοκ για τι τελικέ του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι για τι ε, θερμέ σα ευχαριστίε και τι ε, πρόσδεκτε τροπολογίε σα. Είναι πολλέ παρεμβάσει για να τι σχολιάσω όλες. Το ΝΑΤΟ ήταν ένα θέμα που επανέλθω πολλέ φορέ. Οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή ε, συμφώνησαν να υπάρξει η έκκληση αυτή και καλωσόρισαν την πρόσκληση προς, την, ε, προς το Μαυροβούνιο. Βεβαίω, η Γκουε, το FN της Γαλλίας και η κυρία Λούνατσεκ δεν είναι τόσο ικανοποιημένη με την έκκληση ένταξη προ τον ΝΑΤΟ, αλλά αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, ήταν αμφιλεγόμενο και στις προηγούμενες εκθέσει μου και παρόλα αυτά οι εκθέσει επιβίωσαν. Τώρα, ε, για την ε, κυρία Λούνατσεκ να πω ότι δεν θυμάμαι στο παρελθόν να ήθελε λεπτομερείς ε, τροπολογίες για το ενεργειακό μείγμα του Μαυροβουνίου ή τα προγράμματα ανάπτυξης των υδροηλεκτρικών του δυνατοτήτων, αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα εσωτερικό που ως κυρίαρχο κράτο μπορεί να το αποφασίσει μόνο το, το Μαυροβούνιο. Παραμένοντας βεβαίως ε, συνεπές με το κοινοτικό κεκτημένο. Ούτε εγώ μπορώ να πω στους Μαυροβούνιου να οργανώσουν δημοψήφισμα για τον ΝΑΤΟ. Μόνο το κοινοβούλιο το δικό τους μπορεί να το αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πρόταση στη δική μου τη χώρα. και βεβαίως κάθε χώρα έχει την... Ε, ευθύνη να αποφασίζει μόνη της αν θέλει να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ ή όχι. Κατά τα άλλα τα περισσότερα από τα υπόλοιπα σχόλια νομίζω ότι τα έχω καλύψει. Την καταπολέμηση της διαφορά, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Ο κύριος Καν εκ της κυρίας Ντότζαν έφερε το θέμα των ε, υποκλοπων επίσης ε, η παρέλαση Λουάλ ε, αναφέρθηκε και αυτή. Χαίρομαι που άκουσα από τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή ότι θα γίνει στην Ποντγκόριτσα. Επίση, η κυρία Σουίτσα έκανε σχόλια για τα συνοριακά ζητήματα με την Κροατία και την ατιμορρυσία των εγκλημάτων πολέμου. Θα έλεγα να κοιτάξει την παράγραφο 26 και 27, που νομίζω ότι καλύπτουν και τα δύο αυτά σημεία. Αλλά αν έχει περισσότερα σχόλια να μου κάνει, θα μπορούσε να υποβάλει σχετικά τροπολογίε. Ο νέο εκλογικό νόμο αναφέρθηκε και θετικά, το έχω σχολιάσει και αυτό. Νομίζω λίγο πολύ κάλυψα τα περισσότερα ε, ζητήματα. Ε, το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που πραγματικά είναι μια επιτυχημένη περίπτωση. Τα πάει πολύ καλά, με πολύ καλέ επιδόσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Αυτό αναφέρει και η έκθεσή μου, αλλά βεβαίω και τι διάφορε ελλείψει που παραμένουν στην ολοκλήρωση αυτή τη ευρωπαϊκή πορεία. Όμω αυτή η πορεία για την ώρα είναι από τι πλέον σταθερέ. Να ευχαριστήσω και τέλο και τον κύριο Κούκαν για τα θερμά του λόγια, δεδομένη τη τεράστια πείρα του στην ε, γεωγραφική αυτή ζώνη. Και ε, είναι πολύ σημαντικές οι θετικές ε, κουβέντες από μέρους του ως έμπειρο πολιτικού. Ε, σας ευχαριστώ μέχρι την επόμενη μας συζήτηση. Ευχαριστούμε. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Και έτσι κλείνουμε το σημείο 4. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα προτού περάσουμε σε επόμενο θέμα. Welcome back, ladies and gentlemen. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και πάλι. Προχωρούμε στο θέμα ε, για την Αίγυπτο με τον ε, κύριο Πάτρικ Κοστέλο που είναι επικεφαλής του τμήματος ε, Μέσης Ανατολής που καλύπτει Αίγυπτο, Λίβανο και Ιορδανία. θα μας ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα, καθώς και για τον πολιτικό διάλογο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Με χαρά θα ακούσουμε τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών. Ξέρετε ότι από το 2012 το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου δεν συνεδριάζει. Τώρα για πρώτη φορά έχουν συγχωνευτεί τα δύο κοινοβουλευτικά ε, σώματα. Και η Επιτροπή μας πρόκειται να σκεφτεί την Αίγυπτο στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2016. Εμείς, ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με την αντίστοιχη Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Αιγύπτου και θέλουμε να βοηθήσουμε στη σύσταση Επιτροπών που θα επιτρέψουν την καλύτερη νομοθεσία, ιδιαίτερα στο θέμα της δικαστικής εξουσίας και του κράτους δικαίου. Ιδιαίτερο ε, θέμα είναι το καθεστώς της νομοθεσίας, ε, ιδίως από την άποψη της ε, απουσίας κοινοβουλευτικού σώματος και νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, διαδηλώσεις. Στις 15 και 16 Νοεμβρίου διεξήγαμε μια ε, συζήτηση διεξήχνει συζήτηση της αποστολής στην Αίγυπτο και θα μας ενημερώσει ο κύριος Κοστέλο και θα συζητηθούν αυτά τα θέματα και στην συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Δικαιοσύνη στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Μετά την, ε, την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μογκερίνη στην Αίγυπτο τον Νοέμβριο, όπου συζητήθηκαν ε, ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και η περιφερειακή κατάσταση ε, όσον αφορά τη μετανάστευση και την Λιβύη. Επίσης έθεσε ζητήματα που σχετίζονται με, τη, με τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας με σεβασμό στο κράτος δικαίου. Κύριε Κοστέλο, σας καλωσορίζω, έχετε το λόγο. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλείτε σε αυτήν την Επιτροπή για να σας ενημερώσω και θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό. Οι εκλογές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη ε, στην Αίγυπτο. Υπάρχουν κάποιοι τελικοί ε, ε, ε κύκλοι στις 15 και 16 ε, Δεκεμβρίου. Η δική μας αποστολή αποτελούνταν από τρεις εμπειρογνώμονες και κατέληξε ότι οι εκλογές ήταν πιο πολύ μια διοικητική διαδικασία και όχι τόσο δημόσια. Η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλή ε, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων. Όσον αφορά ε, τις προοπτικές του Κοινοβουλίου, εκλέχτηκαν 120 βουλευτές από τέσσερις εκλογικές περιφέρειες και από εκλογικές λίστες και 548 από ε, μονοεδρικές περιφέρειες. Οι γενικές τάσεις και εδώ αυτό προκύπτει από την εξολόγηση της ε, αποστολής εμπειρογνωμών μας. Η, η οργάνωση των εκλογών δεν ήταν ιδιαίτερα διαφανής και καθώς όπως είπα ο χαρακτήρας των εκλογών ήταν κυρίως διοικητικός οι εκλογικές επιτροπές ε, με επικεφαλής 1.600 δικαστικούς αντιπροσώπους ε, υπήρξε μια πολύ χαμηλή συμμετοχή ιδιαίτερως μεταξύ των νέων ανθρώπων και φαίνεται ότι κυρίως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ψήφισαν καθώς ε, η συμμετοχή ανακοινώθηκε ότι κινήθηκε στο 28%. Οι προεκλογικές εκστρατείες ήταν ανάμικτες. Υπήρξε απαγόρευση ε, να γίνουν εκστρατείες σε τζαμιά, κάτι που δεν ίσχυσε για τις εκκλησίες. Χρησιμοποιήθηκαν και ιδιωτικά κανάλια για να ενισχυθούν συγκεκριμένοι υποψήφοι. Ενώ ο νόμος για, την, για τις διαδηλώσεις ε, όρισε και την κατάσταση στην οποία έπρεπε να κινηθεί η αντιπολίτευση. Ευρύτερα, ο νόμος για τις διαδηλώσεις καθώς και η αντιτρομοκρατική νομοθεσία δημιούργησαν ε, ένα εκλογικό πλαίσιο που δυσχέρανε τη συμμετοχή. Πολλοί ακτιβιστές, αντιπολιτευόμενοι, μέλη νέων, ε, κινημάτων ε, νεολαίας βρίσκονται στη φυλακή. Το Κοινοβούλιο έχει μεταξύ των μελών του πολλούς ε, προεδρικούς υποψήφιους, αλλά και περισσότερες γυναίκες. Γενικά, οι Ισλαμιστές, οι αριστεροί και οι πρώην ε, ε, υποστηρικτές του Μουμπάρακ δεν είχαν επιτυχίες στις εκλογές. Εμείς από την πλευρά μας θα πιέσουμε για να ε, βελτιωθεί η εκλογική νομοθεσία και να ανοίξει ο δημόσιος χώρος και η δημόσια συζήτηση στην ε, Αίγυπτο. Τώρα, η παρουσία του Κοινοβουλίου ε, στην Αίγυπτο είναι ζωτική σημασία προκειμένου η χώρα να κινηθεί σε θετική κατεύθυνση. Όχι μόνο πρέπει να διασφαλιστεί ο έλεγχος εκτελεστικής εξουσίας. Καθώς το, το σύστημα είναι προεδρικό, αλλά θα πρέπει να εξετάσει και ένα νέο σύνταγμα το οποίο υπερψηφίστηκε σε δημοσίευμα το 2014. Αυτό το νέο σύνταγμα διαθέτει μια ε, σειρά από ε, προοδευτικές διατάξεις οι οποίες έχουν υπονομευθεί από την εκτελεστική εξουσία. Το ε, άρθρο 156 του συντάγματος επιτρέπει το, στο Κοινοβούλιο ε, να ε, εντός 14 ημερών να αναπέμψει προεδρικά διατάγματα. Και θα επανέλθω στο ζήτημα του διαλόγου για τα ανθρώπου, ανθρώπινα δικαιώματα ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα να ε, επηρεάσει ή να ε, λάβει απόφαση ε, επί των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν το διάστημα της απουσίας του Κοινοβουλίου. Όπως είπατε για τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Αιγύπτου, η είπατε εκπρόσωπος Μογκερίνη επισκέφθηκε στις 2 Νοεμβρίου το Κάιρο και στη βάση των συναντήσεων που οργανώθηκαν υπήρξε ε, συμφωνία για την επανέναρξη της διαδικασίας Επιτροπής Σύνδεσης και γι' αυτό ε, υπήρξε και ένας πολιτικός διάλογος 15 και 16 Νοεμβρίου ε, στο Κάιρο. Πρόκειται για την πρώτη υποεπιτροπή εδώ και πέντε χρόνια που συστήνεται με τους Αιγύπτιους ε, για πολιτικά ζητήματα. Είναι σημαντικό το βήμα αυτό λοιπόν. Αναφερθήκατε στο ζήτημα διαφόρων ε, νομοθετικών πράξεων. Να σας δώσω μια εικόνα για τα ζητήματα που θέσαμε στον διάλογο για τα πολιτικά ζητήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους Αιγύπτιους. Είπαμε ότι ο νόμος 107 ε, πρέπει να καταργηθεί ο νόμος για τις διαδηλώσεις. Και θα πρέπει ο νόμος 914 ε, ε, για τις συναθρήσεις να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει επίσης να απελευθερωθούν όλοι όσοι έχουν φυλακιστεί στη βάση του νόμου αυτού. Επίσης, ζητήσαμε την ανάκληση του άρθρου 78 ε, του ποινικού κώδικα για την ε, χρηματοδότηση από το εξωτερικό πράξεων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας. Επίσης πρέπει να ε, αντικατασταθεί ο ε, νόμος και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα. Η Αίγυπτος σημείωσε ότι ε, προετοιμάζεται νέα νομοθεσία αλλά συνεχίζει να θέλει να ελέγχει την χρηματοδότηση Κατηγορηθήκαμε δε ότι ε, διαταράσσουμε τις σχέσεις της κυβέρνησης με την κοινωνία των ε, πολιτών. Εμείς επίσης αναφερθήκαμε στην κατάχρηση του ποινικού κώδικα και στο άρθρο 102 όσον αφορά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι Αιγύπτιοι τόνισαν ότι υπάρχει ε, σε εξέλιξη μια δημοκρατική μεταρρύθμιση με ε, ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου και ε, ομολόγησαν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από το Κοινοβούλιο αλλά χρειάζεται και αναθεώρηση του συντάγματος για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Ένωση και η Αίγυπτος εξετάζουν το ζήτημα της ταχύτητας των μεταρρυθμίσεων με διαφορετικό τρόπο, αλλά υπάρχουν περιθώρια και θα τα αξιοποιήσουμε. Έχουμε πλέον μια συμφωνία την οποία θα εξετάσουμε σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή αλλά και άλλες ε, υποεπιτροπές που θα ε, συνεδριάσουν τους επόμενους μήνες. Επίσης, παράλληλα με τη διαδικασία πολιτικού ε, διαλόγου υιοθετήθηκε και η διαδικασία ε, καλής γειτονίας στην Ευρώπη με προσαρμοσμένη προς κάθε χώρα προσέγγιση. Έπειτα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα υιοθετήσει συμπεράσματα για το θέμα αυτό θα αρχίσουμε συνομιλίες με τους Αιγύπτιους για το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Δεύτερο σημείο. Μία από τις προτεραιότητες στον προγραμματισμό μας ε, όσον αφορά την χρηματοδοτική στήριξη της Αιγύπτου αφορά τη διακυβέρνηση και επαναρχόμενος σε αυτό που είπα για την ανάγκη συνεργασίας και ενίχυσης του Κοινοβουλίου προφανώς αυτό θα αποτελέσει μια από, ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας. Τέλος θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι Όσο η είπατε εκπρόσωπος ήταν στο Κάιρο, εκφώνησε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο της πόλης και ένα από τα ζητήματα τα οποία ε, ανέδειξε ήταν το γεγονός ότι η μέση ηλικία στην Αίγυπτο είναι τα 25 χρόνια. Σε μια χώρα 60 εκατομμύριων αυτό ε, αποτελεί μια, μια τεράστια δυνατότητα για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η χαμηλή συμμετοχή λοιπόν στις εκλογές, και ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό που είπε είναι ότι αν δεν ε, δημιουργήσουμε ένα μέλλον για τους νέους ανθρώπους ενδεχομένως αυτοί να στραφούν σε εκείνους που υπόσχονται διάφορες εναλλακτικές άρα θα πρέπει ε, και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αύξηση του βιωτικού επίπεδου να είναι ένας που καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την ε, δραστηριότητά μας και τη συμμετοχή μας, την βοήθειά μας προς την Αίγυπτο. Ε, είμαστε πολύ σαφείς όσον αφορά τις διαφωνίες που έχουμε με τη χώρα για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα ζητήματα που έχει θέσει και το Ευρωκοινοβούλιο πολλές φορές και με στεναρότητα, αλλά υπάρχει ε, ανάγκη να στηριχθούν οικονομικά οι άνθρωποι στην Αίγυπτο προκειμένου να... διότι ε, το βιωτικό επίπεδο ε, αν δεν αυξηθεί έχει τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στο μέλλον για τη χώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Παντσέρη. Ε, Ευχαριστώ. Είναι εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το υπογραφήσουμε. Η Αίγυπτος έχει στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην όλη περιοχή. Οπότε είναι και σκόπιμος και επιβαλόμενος ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου για να αναθερμαθούν οι σχέσεις μας. Πρέπει να πω όμως ότι αυτά που άκουσα από τον κύριο Κοστέλο διαγράφουν μια κατάσταση αρκετά προβληματική από πολιτική σκοπιάς και ως προς το τι συμβαίνει με τα δικαιώματα. Η έντονη αίσθηση που αποκομίζουμε είναι ότι στη δίκαιη μάχη κατά της τρομοκρατίας στην πραγματικότητα πολλές φορές αυτό, αυτή η μάχη χρησιμοποιείται ως άλοθη για να περάσουν ε, πολιτικές καταστολής των δικαιωμάτων. Έτσι δυσκολεύεται και η Ευρώπη να δώσει τις σωστές ενδείξεις. Διότι αν διαβάσει κανεί σήμερα τις εφημερίδες θα δει ότι Στη Γαλλία εδώ γίνεται μια συζήτηση για προσωρινή φυλάκιση των υποποπτών για τρομοκρατία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για χιλιάδες άτομα και μιλάμε και για συνέπεια πολλές φορές το τι συμβαίνει στην πράξη. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της απόλυτης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της ασφάλειας και άμυνας από την άλλη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Αίγυπτος να ε, αποκλίνει από τη θετική κάλυψη των προστατευτικών δικαιωμάτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και με όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στις διάφορες ε, διαδηλώσεις. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό θα είναι η τελευταία μου παρατήρηση, η ομιλία της κυρίας Μογκερίνη στο Κάιρο να είναι ένας καλός ιονός σε σχέση με την ομιλία του Ομπάμα στο Πανεπιστήμιο του Καϊρού. Να αρχίσει δηλαδή να ανοίξει μια νέα προοπτική για την μεσογειακή προοπτική της χώρας αυτής σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη, πολύ δυσχερή και ελπίζω να μας φέρει τύχη η ομιλία της κυρίας Μογκερίνη στο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Uh, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εστερνιστώ μερικά σχόλια του κυρίου Παντζέρη, γιατί σίγουρα είναι ε, ηγετική αραβική χώρα η Αίγυπτος με ζωτικό γεωστρατηγικό ρόλο και πολλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε με θετικό τρόπο αυτή τη χώρα και να στηρίξουμε αμέριστα την προσπάθειά της. Γιατί Ιδιαίτερα στη χερσόνηση του Σινά υφίσταται τεράστιες ε, τρομοκρατικές απειλές. Είδαμε την κατάληψη ρωσικού αεροπλάνου στο... που απογειώθηκε από το Σάρμελ Σέικ. Φαίνεται ότι το Ισλαμικό κράτος έχει παρισφρήσει και στην Αίγυπτο και φυσικά ε, το ρόλο τους, ε, των αδερφών μουσουλμάνων του Μόρση. Σίγουρα χαιρετίζουμε την προσπάθεια της κυρίας Μογκερίνη και την επίσκεψή της εκεί και χαίρομαι που ξεκίνησε και πάλι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αίγυπτο. Σίγουρα το βασικό μήνυμα της κυρίας Μαγκερίνη ήταν η ανάγκη να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να δοθούν προοπτικές για τους νέους στην Αίγυπτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεδομένου ότι 25% είναι ο μέσος όρος ηλικίας στην Πολύ αυτή η χώρα. Τώρα, ε, ε, έχουμε, είχαμε το δεύτερο γύρο των εκλογών και όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μεγάλο το ποσοστό αποχής. Κρίμα που ιδιαίτερα οι νέοι ε, μποϊκοτάρισαν τις εκλογές. Βέβαια χαίρομαι γιατί εξελέγησαν περισσότερες γυναίκες και οι μεγάλοι τιμένοι ήταν οι Ισλαμιστές και οι Σαλαφιστές. Οπότε σίγουρα θα έχουμε μια πιο ανεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και πιο κοσμική, λαϊκή Αίγυπτο. Βέβαια έχουμε το άρθρο 156 που δίνει ιδιαίτερες ε, εξουσίες στον πρόεδρο γιατί είναι σχεδόν ημιπροεδρικό το σύστημα. Γι' αυτό και παρακολουθούμε ενδιαφέρον και θα το νέο κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Πάντως ε, η ομάδα ECR είναι ε, στενός φίλος της Αιγύπτου και μάλιστα ε, ως μέλος της ε, ομάδας των φίλων της Αιγύπτου περιμένω με ανυπομονησία την επίσκεψή μας στη χώρα αυτή του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαμπάλεν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία η κίνηση της Αιγύπτου προς περισσότερη σταθερότητα να τύχει της υποστήριξης της δύση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αν ανατραπεί η σταθερότητα της Αιγύπτου δεν θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την προσφυγική κρίση ή την επέλαση του Ισλαμικού κράτους. Χρειαζόμαστε ανοιχτό διάλογο με την Αίγυπτο και θα ήθελα η αντιπροσωπεία να μου πει αν η νεοεκλεγήσα Αιγυπτιακή Βουλή θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής ή μήπω είναι ένα κοινοβούλιο ίσονος σημασίας. Ευχαριστώ κύριο Σαφόιζερ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ιστορική υπενθύμηση στους συναδέλφους. Ποιος ε, στήριξε την Αραβική Άνοιξη, ποιος έβαλε στην εξουσία τους σαλαφιστές και τους αδερφούς μουσουλμάνους, ποιος ε, μάλιστα και πρόσφατα δεν στήριξε τον πρόεδρο Σίση και ο προσ, προσπάθησαν να, να δολοφονήσουν και τον πρόεδρο. Ε, το ξέρετε θαυμάσια όλοι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν αυτέ. υπεύθυνε για όλη αυτή την κατάσταση. Και πάλι έχουμε μία απόπειρα αποσταθεροποίηση που ευτυχώ ε, πέτυχε. Γιατί αν είχε τελεσφορήσει αυτή η απόπειρα σταθεροποίηση, ε, η κατάσταση στην Ευρώπη θα ήταν ακόμη χειρότερη. Οπότε αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξει αυτή την κοσμική λαϊκή κυβέρνηση, τη ρεπουμπλικάνικη κυβέρνηση της Αιγύπτου, που συνεχίζει να είναι βαθύτατα μουσουλμανική, είναι πολύ θετικό. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε τον πρόεδρο Σίση, γιατί διακυβεύεται και η δική μας επιβίωση. Αν αποτύχει ο πρόεδρος Σίση, θα αποσταθεροποιηθεί πλήρως ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μιας δικής του αποσταθεροποίησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την ενημέρωση για το, τα γεγονότα στην Αίγυπτο. Και συμμερίζομαι και εγώ το σχόλιο του κυρίου Παντσέρη. Να μην ξεχνούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σίγουρα η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική χώρα όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω της επιρροής της στον αραβικό κόσμο. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο για περισσότερο διάλογο με την Αίγυπτο. Φυσικά θα πρέπει και η Αιγυπτιακή Βουλή να θέσει καλύτερες προδιαγραφές όχι μόνο για τον Αιγυπτιακό λαό, αλλά και γενικότερα για τον Αραβικό κόσμο. Γιατί όλοι προσβλέπουμε στη σταθερότητα και στην ασφάλεια. Αλλά ποτέ μια δικτατορία δεν θα εξασφαλίσουν σταθερότητα και ασφάλεια. Γιατί είναι μετρημένα, μετρημένες ημέρες τέτοιων καθεστώτων. Χαίρομαι για την εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα, αλλά μας είπατε ότι ήταν μεγάλη αποχή και μάλιστα η αποχή κυρίως των νέων. Οι νέοι είναι το μέλλον της Αιγύπτου και οι νέοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αν δεν έχουμε νομοποίηση και σταθερότητα, τι θα γίνει. Μας ανησυχεί η βία που επικρατεί στην χώρα αυτή και η τρομοκρατία. Και σίγουρα αν απαγορεύουν τα τζαμιά αλλά όχι και τις εκκλησίες, ουσιαστικά ρίχνουν νερό στο μήλο των τρομοκρατών. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ίση, ισότιμη μεταχείριση. Αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε αξιόπιστο αφήγημα. Μακάρι να σταθεροποιηθεί η Αίγυπτος, γιατί και εγώ θα ήθελα να γίνει σταθερή και ισχυρή χώρα και να διαδραματίσει θετικό ρόλο. Ευχαριστώ. Κύριε Κοστέλο, πριν σας ξαναδώσω το λόγο, έχω μια σύντομη ερώτηση. Στην ενημέρωσή σας δεν αναφέρατε καθόλου τους χριστιανούς τις χριστιανικές κοινότητες. Οι χριστιανοί είναι η θρησκευτική μειονότητα που έχει υποστεί τους μεγαλύτερους διωγμούς στην περιοχή. Πώς να εκλάβω την παράληψη αυτή. Να θεωρήσω ότι η κατάσταση των χριστιανών στην Αίγυπτο είναι άψογη. Ή υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτή την παράληψη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να σχολιάσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια και τις απόψεις που εκφράστηκαν. Θεωρώ ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συμφωνούμε όλοι εδώ μέσα για την στρατηγική σημασία της Αιγύπτου τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ωστόσο διάφορες ε, αποχρώσεις που εκφράστηκαν από τους ε, βουλευτές. Μια σκέψη για το ζήτημα της σταθερότητας και της δημοκρατίας, θα ήθελα να πω. Πολλές φορές αυτό το θέμα τίθεται ως ε, θέμα επιλογής. Εμείς θεωρούμε ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι φυσικά πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε την Αίγυπτο στο δρόμο της προς την σταθερότητα και αυτό ακριβώς είπε και η κυρία Μογκερίνη στην επίσκεψή της στο ΚΑΕΡΟ. αλλά ο λόγος για τον οποίο θέτουμε το ζήτημα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάγκης αλλαγής τροποποίησης των νόμων για την ενίσχυση της συμμετοχής είναι διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας από τους τρόπους για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια σταθερότητα και η ε, καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στην Αίγυπτο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ε, ενεργότερης ε, εμπλοκής μας με τη χώρα αφενός και αφετέρου στο να καταστήσουμε σαφές ότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και να κάνουμε βεβαίως και ό,τι μπορούμε μέσω της, ε, του έργου της διακυβέρνησής μας για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Για το ζήτημα των χριστιανών, ε, νομίζω ότι είπα ότι οι προεκλογικές εκστρατείες απαγορεύτηκαν στα τζαμιά αλλά όχι στις εκκλησίες. Κάτι που αντικατοπτρίζει και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε σύγκριση με ό,τι ε, συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια. Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην ε, συνάδελφό μου τη Λόρα Μπορίσοβα, που είναι αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος για τις Εκλογές. Ευχαριστώ να συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Έχουμε επιδείξει ε, την προθυμία μας να στείλουμε μια ε, πλήρη ε, αποστολή παρατηρητών για τις εκλογές και μια μικρότερη φέτος. Υπήρξαν κάποιες συστάσεις που δημοσιεύτηκαν πέρσι έπειτα από αυτή την αποστολή την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε. Θα επαναληφθούν αυτές στην ε, αποστολή εμπειρογνωμόνων αυτή τη μικρότερη ομάδα που επισκέφθηκε την ε, χώρα φέτος. Ε, εξετάζουμε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εκλογική νομοθεσία στην Αίγυπτο. Εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους η συμμετοχή ήταν χαμηλή. Ενδεχομένω εκτός από νομικούς, εκτός από τους πολιτικούς λόγους υπήρχαν και νομικοί λόγοι. Θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά προκειμένου να συνεργαστούμε και με τους Αιγύπτιους εταίρους μας εν ώψη και των τοπικών εκλογών που θα διοργανωθούν την επόμενη χρονιά προκειμένου να αυξηθεί και να ενισχυθεί η διαφάνεια στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ε, χρονοδιάγραμμα ε, για την εκδίκαση των ενστάσεων που ε, υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή. Υπήρξαν πολλές τέτοιες ενστάσεις ε, στις φετινές εκλογές. Αυτό βεβαίως δημιουργεί μια αβεβαιότητα και όλα αυτά τα μέτρα είναι ε, ζητήματα τα οποία, όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία θέλουμε βεβαίως να συζητήσουμε με τους εταίρους μας. Να πω, ε, γιατί ξέχασα να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα του κ. Βαμπάλινς για το πώς το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο θα ε, συμπεριφερθεί, ποια θα είναι η θέση του ε, και η σχέση του με την κυβέρνηση. Ε, φυσικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει έως ότου συσταθεί σε σώμα το Κοινοβούλιο. Ε, θεωρούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει, η έκβαση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Αφενός βεβαίως από, την, από τον πολιτικό συσχετισμό εντός του Κοινοβουλίου, αφετέρου από το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να εργαστεί το Κοινοβούλιο και τρίτον από το κατά πόσο άλλοι, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν το Κοινοβούλιο στις εργασίες του. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ε, το πράγμα τα, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Κοστέλο. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο. Σημείο 6. Ενημέρωση για τις, κοινοβουλευτικές, ε, για τις βουλευτικές εκλογές ε, στο Μιανμάρ που έγιναν στις 6 Νοεμβρίου του 2015 ενημέρωση από την επικεφαλής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας παρατήρηση των εκλογών. Επαναλαμβάνω, ε, το Κοινοβούλιο έστειλε αντιπροσωπεία παρατήρηση εκλογών για τις βουλευτικές εκλογές της Μιανμάρ που έγιναν, έλαβαν χώρα στις 8 Νοεμβρίου. Έγιναν μάλιστα σε φιλελληνική ατμόσφαιρα και το κόμμα της Αν Σαν Σουκί, το NLD, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία, ε, ε, κέρδισε συντριπτική νίκη με 80% των βουλευτικών εδρών. Και παράλληλα το γεγονός 25, ότι 25% των βουλευτικών εδρών του Κοινοβουλίου προορίζονται για το στρατό, μετά τις εκλογές, το κόμμα NLD της Σαν έχει μια σαφή απόλυτη πλειοψηφία, 60% στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου της Μιανμάρ. Το USDP, το Φιλοστρατιωτικό Κόμμα, είναι το δεύτερο κόμμα του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Βέβαια, με βάση το Σύνταγμα, η Άνσαν Ξουκή αποκλείεται από την Προεδρία, ε, αλλά απεφάνθη ότι όποιο και είναι ο Πρωθυπουργό, ε, ο Πρόεδρο θα κρατήσει εκείνη τα ενία των αποφάσεων και τη εξουσία ε, ω ε, Πρόεδρο του κόμματό τη. Πάντω ήταν σημαντικές εκλογές, επικεφαλή της κοινοβουλευτική αντιπροσωπής των ο κύριος και θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ήδη ποια ήταν τα αποτελέσματα και ποιε οι παρατηρήσει μα την ημέρα των εκλογών. Είναι σημαντικό πάντως να αναγνωρίσουμε ότι οι εκλογές αυτές σε μία χρονιά που έχουμε πολλές κρίσεις, πολλά δυσάρεστα μαντάτα και πολλά προβλήματα, ίσως ήταν μία πολύ θετική νότα και μία ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Η χώρα απέκτησε νέο σύνταγμα το 2008, δημιουργώντας έτσι τις ε, προϋποθέσεις ε, ή κάποιες προϋποθέσεις για τις εκλογές. Όπως είπατε όμως 25% ε, και στην Άνω και στην Καταβουλή των εδρών ε, προορίζονται για το στρατό και καθορίζονται από το, από το Γενικό Επιτελείο. Αυτό είναι μια επαναχώρηση βέβαια σε ένα κανονικό και δημοκρατικό εκλογικό πλαίσιο. Το 2010 έγιναν γενικές εκλογές, στις οποίε μποϊκοτάριξε το κόμμα της Αν Το 2011 ξεκίνησε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων ε, που διήρκεσε και το 2012. Έγιναν οι πρώτες εκλογές και σε 40 εκλογικές περιφέρειες το NLD ε, κέρδισε συντριπτική νίκη. Βέβαια, ε, για τις εκλογές της 8 Νοεμβρίου Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις γιατί διαπιστώθηκαν πολλά τροτά σημεία και πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα το νομικό πλαίσιο δεν ήταν καθόλου ιδεώδες. Δεύτερον, η Επιτροπή των Εκλογών δεν είχε εμπειρία για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό φάνηκε. Υπήρχαν αρκετέ αδυναμίε. Ούτε υπήρχε σαφήνεια για το κατά πόσο η αρμόδιες αρχές θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και ανοιχτών εκλογών και αν το επέτρεπαν αν θα σέβονταν τα αποτελέσματα, την έκβαση των εκλογών. Όλα αυτά ήταν ασαφή πριν τις εκλογές. Επίσης ε, κάποια τμήματα της χώρας ε, είχαν χτυπηθεί από θεομηνίες, από ε, βία μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων Υπήρχαν διάφορα τροτά σημεία, όπως σας είπα, πριν τις εκλογές και προσθέθηκα και κάποια σημεία ειδικά που σχετιζόταν με τις εκλογές. Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα ηλεκτρονικό αρχείο από την Εθνική Εκλογική Επιτροπή και υπήρχε πρόβλημα αν θα ε, είναι πλήρης αυτός ο ψηφιακός κατάλογος και το θέμα το κατά πόσο ήταν ελεύθερες οι προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων, γιατί υπήρχε περιορισμοί στο δικαίωμα του, συν, του συναθρίζεστε, του συνέρχεστε. Επίσης, δημιουργήθηκε και ένα ριζοσπαστικό βουδιστικό κίνημα, κάτι που ακούγεται αντιφατικό ριζοσπαστικό και βουδιστικό. Είναι ένα ριζοσπαστικό, εθνικιστικό, ε, βουδιστικό κίνημα που ε, τάχθηκε υπέρ της ε, θέσπισης τεσσάρων νομοθετημάτων, υπέρ της προστασίας της εθνικής και της κριτικής ταυτότητας. Πάντως, παρά τις αδυναμίες αυτές, ήταν αξιοσημείωτη η πρόσκληση ε, των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την παρακολούθηση αυτών των εκλογών. Ήμουν επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας ε, και πριν περάσω στις παρατηρήσεις της αντιπροσωπείας μας, θα ήθελα να πω ότι στην αποστολή αυτή παρατηρήσαμε μια αγαστή συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων. Το είπα και στην Ολομέλεια, το επαναλαμβάνω και εδώ και η αντιπροσωπεία μας και, τα και το FBI και η αποστολή παρατήρησης ε, εκλογών δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ούτε τα κράτη-μέλη τη Δευτέρα μέσα μετά τις εκλογές ε, δεν εξέδωσαν ανακοινωθέντα τύπου, αλλά κράτησαν την ε, διακριτικότητα και τη σιωπή που ήταν απαραίτητη, γιατί συνήθως τα αποτελέσματα βγαίνουν ολοκληρωμένα δύο μέρες μετά τις εκλογές. Η προσέλευση ήταν ε, σχετικά ενθαρρυντική, υπήρχε ανταγωνιστικότητα, υπήρχε φιλιρινική διεξαγωγή, ήταν ε, γύρω στο 70% η προσέλευση στις κάλπες. Και πραγματικά ήταν συντριπτική η νίκη του, του κόμματος της Σαν Σουκί, του NLD. Τα εκλογικά αποτελέσματα έγιναν δεκτά με ψυχραιμία, με ηρεμία και ε, ήταν σημαντικό ότι το, οι τυθέντες των εκλογών αποδέχτηκαν τα αποτελέσματα και μερικές φορές η συμπεριφορά των νικημένων είναι πιο σημαντική από τη συμπεριφορά των νικητών σε τέτοιες εκλογές. Το USDP δέχτηκε την δημοκρατική ήττα στις εκλογές και παρότεινε και τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία στην όλη εικόνα που είναι πιο δύσκολα. Το 25% των εδρών, όπως σας είπα, προορίζεται στο στρατό. Και το NLD, παρόλο που έχει 80% των ψήφων, μόνο το 60% των εδρών δικαιούται στις δύο βουλές. Επίσης, δεν θα υπάρξει ούτε ένας μουσουλμάνος εκπρόσωπος στη Βουλή. Σε μια χώρα, μάλιστα, που έχει μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα. 5 έως 10% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, αλλά δεν θα έχουν ούτε ένα βουλευτή. Και πολλοί στερήθηκαν τα δικαιώματά τους. Αυτό στυλιτεύτηκε από πολλούς. Επίσης το θέμα της επικότητας. Άνθρωποι που ήταν ε, πρώην βουλευτές δεν μπόρεσαν να επανεκλεγούν γιατί δεν μπορούσαν να αποδείξουν ε, ότι και οι διαγωνιστές τους ήταν ε, υπήκοοι Μιανμάρ. Πάντως ήταν γενικώ θετικά τα αποτελέσματα. Τώρα για το μέλλον. Τι γίνεται πέραν της εκλογικής διαδικασίας. Το σαφές είναι ότι ο λαός της Μιανμάρ ψήφισε για αλλαγή και περιμένει την αλλαγή. Οπότε η διαχείριση της ε, μετάβασης ε, θα είναι πολύ σημαντική πρόκληση. Ο πρόεδρος του RLD συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με τον ε, αρχηγό Γεθά για να συζητήσει αυτές τις αλλαγές. Το κόμμα CommonLD βέβαια δεν έχει μεγάλη πείρα στην ηγεσία. Αυτό είναι διαπίστωση, δεν είναι καμία κριτική. Δεν έχει ιδιαίτερο εκλογικό πρόγραμμα, δεν έχει πλατφόρμα, δεν έχει διεξοδικές απόψεις για τους διάφορους τομείς. Και παρόλο ε, η μουσουλμανική μειονότητα η Μποχήμ ε, στερήθηκε τα εκλογικά δικαιώματα, η Μιαμάρ είχε και άλλες μειονότητες. Και το NLD κέρδισε ε, ψήφους και σε Περιοχέ με σημαντική εθνοτική παρουσία άλλων μειονοτήτων και ίσω αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται αρκετά. Και παρά την αλλαγή, ο στρατό εξακολουθεί να κατέχει το δικαίωμα άρνηση για τη μεταρρύθμιση του συντάγματο, για την αναθεώρηση του συντάγματο αυτό το 25% των εδρών που κατέχει. Τώρα, θα υποβάλω την τελική μου έκθεση στα τέλη Μαρτίου θα περιλαμβάνει αρκετά συμπεράσματα. Καταρχήν το 25% των εδρών για το στρατό. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις διεθνείς προδιαγραφές της δημοκρατίας. Περιορισμοί στο δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν. Επίσης, οι περιορισμοί για τον υποψήφιο στην Προεδρία. Δεν μπορεί κάποιο να είναι υποψήφιο για πρόεδρο συνταγματικά εφόσον ο σύζυγο ή τα τέκνη και τα δύο είναι αλλοδαπιπολίτε. Αυτό είναι άνευ προηγουμένο. Πρωτοφανέ για μια χώρα. Γι' αυτό και υπόκειται σε αυτό το συνταγματικό αποκλεισμό η Αν Σανξουκή. Υπάρχει το πρόβλημα της μετάβασης με τη συνταγματική κατάσταση και την πολιτική κατάσταση που εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πάντως μέχρι στιγμής και οι εκλογές και οι πρώτες συνομιλίε που έγιναν για την επερχόμενη μετάβαση μας δίνουν ε, λόγους ε, για αισιοδοξία και ελπίδα ότι η χώρα θα ακολουθήσει τη σωστή πορεία. Ευχαριστώ και με στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος τώρα στην Ένα που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου σε αυτή την επίσκεψη. Ναι, και ήταν προνόμιο με τους συμμετέχοντες συναδέλφους να είμαι αυτή τη αποστολή. Υπήρχε μεγάλη διάθεση για συμμετοχή και πολύ καλή συνεργασία με τον Αλεξάνδρ Λάμπστορφ. Θα συμφωνήσω απολύτω με όσα είπε, πήγε πολύ καλά η αποστολή, διότι πραγματικά είχαμε όλη την απαραίτητη στήριξη, όχι μόνο από του συνεργάτε του Κοινοβουλίου, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, επιτόπου αντιπροσωπεία μα, όπου πρέπει να ε, σημειώσω ότι είναι πολύ νεαρή, έχει ηλικία μόλις δύο ετών και σε ένα σκηνικό αρκετά κρίσιμο. Δηλαδή μπορέσαμε να έρθουμε σε άμεση επαφή με τους διάφορους εταίρους και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η μέρα των εκλογών πήγε πολύ καλά. Κάποιοι από εμά είπαν ότι ήταν από τι καλύτερες εκλογέ που είχαμε παρακολουθήσει, αλλά υπήρχαν έρευνε και από πριν, τις ανέφερε και ο Αλεξάνδερ, κυρίως με την ε, προσέλευση των ε, μουσουλμάνων ψηφοφόρων, την ε, στέρηση λοιπόν δικαιωμάτων εκλογικών από κάποιους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, τις γυναίκες σε κάποια μέρη της χώρας, και βεβαίω κάποιε δυσκολίε στην ε, διαδικασία καταμέτρηση λόγω τη απειρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν ανεξάρτητε οι εκλογέ ε, και τελικά όλα πήγαν καλά στο τέλο και πρέπει να τονίσω τον εξαιρετικό ρόλο των γυναικών. Όπω είπε και ο Αλεξάνδρ, μόνο 10% γυναικών εξελέγησαν, αλλά έπαιξαν ζωτικό ρόλο σε αυτέ τι εκλογέ, διότι η πλειονότητα των υπαλλήλων ήταν γυναίκε οι περισσότεροι εκπρόσωποι των κομμάτων ήταν γυναίκες, οι επιτόπιοι παρατηρητές ήταν επίσης γυναίκες και είχαν άρτιστη κατάρτιση. Άριστη κατάρτιση. αυτό έδειξε τον εθνικό χαρακτήρα των ανθρώπων της Μιανμάρ, το πόσο συγκρατημένοι μπορεί να είναι και πόσο αξιοπρεπής, αλλά και λόγω της ταυτοτικής νοοτροπίας που επικρατεί μέρη στη χώρα. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια εύρυθμη διαδικασία, διότι τα εκλογικά κέντρα είχαν ε, οργανωθεί με τον ίδιο τρόπο παντού, λειτουργούσαν πολύ καλά και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε επίσης ο Αλεξάνδερ. Τι έγινε με τους ιτημένους και την αντίδρασή τους με τέτοια συντριπτική νίκη η οποία αναμενόταν και επιβεβαιώθηκε. Ήταν επίσης πολύ θετικά τα μηνύματα από εκεί. Ε, πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι η διαδικασία αυτή μετάβασης στην ε, Μιανμάρ είναι κάτι που το περιμένουν πολύ και το ελέγχει ο στρατός με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι θα έλεγα πολύ ισχυρό θεσμό στη χώρα, διότι εκεί είναι κυβερνούσανος τώρα. Και γιατί αυτή η αλλαγή, γιατί αυτή η μετάβαση. Υπάρχει στρατηγικός επαναπροσανατολισμός της χώρας εν ώψη των ε, τόσο δυσβάσταχτων γειτόνων όπως η Κίνα και αναζητούν συμμάχους αλλού. Υπ' αυτήν την έννοια και πέραν των εκλογών Νομίζω εμείς ως Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ανταποκριθήκαμε σωστά με ταχύτητα στη σωστή κατεύθυνση. Κάναμε αυτά που πρέπει. Αναλάβαμε τις πρωτοβουλίες μας για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στην διαδικασία παρατήρηση των εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, που θα είναι και των υστέρων παρακολούθηση. Επίσης, να μην ξεχνάμε τη συμβολή της Αργεντίνη, η οποία μετά την αποστολή είδε ανθρώπους από τη Μιανμάρ που μπορεί να αγωνίζονται σε ε, ένοπλες ομάδες σε άλλες γειτονικέ χώρες ή να βρίσκονται εκεί ως άσυλο ή πρόσφυγες. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με την εθνική συμφιλίωση στη Μιανμάρ και τη διαδικασία τήρησης τη ειρήνη που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ή άλλως. Είναι μεγάλη λοιπόν πρόκληση διότι θα είναι θέμα για τη δημοκρατική διακυβέρνηση τη χώρα στη συνέχεια. Και όλος ιδιαίτερο εν ώψη των πολύ ανησυχητικών τάσεων που ανέφερε ο Αλεξάνδερ, ενό ε, πάρα πολύ αρνητικού, ξενοφοβικού τμήματο ε, θρησκευτικού εθνοτισμού λόγω αυτών των ε, εξτρεμιστών βουδιστών οι οποίοι έχουν κάποιες διασυνδέσεις και με τους κυβερνώντες διαιτητικούς. Βεβαίω, συνταγματική αλλαγή θα χρειαστεί, γιατί το 2008 το σύνταγμα που εγκρίθηκε είναι τελείω ασύμβατο με την δημοκρατία. 25% των εδρών ε, προβλέπονται για το στρατό και επίση ένα μεγάλο ποσοστό τη διακυβέρνηση τη χώρα. Είναι τελείω ασύμβατο αυτό με δημοκρατικό καθεστώ. Όμω, εφόσον ε, κέρδισε με τέτοιο συντριπτικό τρόπο το LND, το ζήτημα είναι αν θα φανούν στο ύψο των περιστάσεων. Για την ώρα δεν είναι ακόμη καν σωστά διοργανωμένη. Δεν υπάρχει απαραίτητη δομή. Υπάρχει Ανσουκή με τους συμβούλους της και μετά υπάρχει ε, ένα πλήθος ε, ταλαντούχων νέων αλλά υπάρχουν τυφωτός απόστασης μεταξύ τους για το μέλλον λοιπόν και να υπογραμμίσω εδώ την μεγάλη σημασία της συμβολής ενός άλλου μέλους της ομάδας μας, της Judith Σαρχεντίνη, η οποία παρακολούθησε και έχει ασχοληθεί με το σχέδιο δημοκρατισμό της χώρας μέχρι τις εκλογές πολύ επισταμένος. Έκανε λοιπόν πολύ συγκεκριμένε προσπάθειες και συνεισφορές για να δει που μπορεί να είναι η δράση μας σκόπιμο και χρήσιμη. Και πάνω από όλα το σημαντικότερο είναι η οικοδόμηση δυνατήτων για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, μεταξύ των οποίων και η διακυβέρνηση των κομμάτων έσω κομματικά και κυρίως του LND που θα είναι το κυβερνών πολιτικό κόμμα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε τι θα πει, πρέπει να καταλάβουν εκείνοι τι θα πει να λειτουργούν σε ένα δημοκρατικό καθεστώ, με την αντιπολίτευση επίσης να λειτουργεί και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους, τι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το καθεξής. Να πω ότι στη συνέντευξη τύπου μας ε, έθεσε ένα θέμα που ξεπερνά το θέμα των εκλογών, όπως είπε και ο Αλεξάνδρ, αλλά αφορούσε και το θέμα των εκλογών, δηλαδή τη στέρηση δικαιωμάτων από τους μουσουλμάνους και το κατά πόσον θα μπορούν να ενταχθούν σωστά οι ε, μειονότητες, οι εθνικές μειονότητες όπως η Ροχίγκα, οι οποίοι δεν ε, συμμετέχουν πλήρως, δεν έχουν όλα τους τα δικαιώματα και δεν τους τα το LND. Εφόσον λοιπόν αυτό το κόμμα θέλει να είναι δημοκρατικό και να ε, εξασφαλίσει τη δημοκρατική διακυβέρνηση, θα πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και σε σύγκριση με τον στρατό που κυβέρνησε τη χώρα ως τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Οπότε να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά παρακαλώ να είστε στο δυνατόν συντομότεροι. Ο κύριος Πλένκοβιτ. Ευχαριστώ για την ε, ενημέρωση Άννα για τις ε, εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μιαμάρ τον Οκτώβριο. Είμαι ο μόνος εκπρόσωπος του ΕΛΚ ε, και θα τοποθετηθώ εκ μέρους των ε, τριών συναδέλφων που συμμετείχαν στην αποστολή παρατηρητών και θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν υψηλή και οι εκλογές οργανώθηκαν ε, καλώς. Ε, δυστυχώς ωστόσο ένα κόμμα που ε, κατακτά το 81% των ε, ψήφων έχει μόνο το 60% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ε, τερματιστούν επιτέλους τα προνόμια του στρατού. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας στην Μιανμάρ και θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η ε, δικτατορία 50 χρόνων στην ε, Μιανμάρ έχει αφήσει τη χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις υποδομές, δεν υπάρχει λιμάνι βαθέως ε, ε, ε, μεγάλου βάθους, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Πολλοί νέοι από την ε, Μιανμάρ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσουν το νέο εκλεγέν κοινοβούλιο να προχωρήσει στο έργο του και να συνάψει και ένα σύστημα συνεργασίας όπως υπάρχει με άλλες χώρες. ευχαριστώ. Θα είμαι ταχιστός διότι συμφωνώ με την ε, παρουσίαση που μας έκανε ο Αλεξάντερ και η συνάδελφος Γκόμες. Είναι η πρώτη φορά που... Είναι η πρώτη φορά που συμμετάσχω σε μια τέτοια αντιπροσωπεία παρατήρηση εκλογών και ήταν μια εμπειρία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται και στην επικεφαλή της αντιπροσωπείας μας, την κυρία Γκόμες, η οποία εργάστηκε υπέροχα με τόσες δεσμεύσεις που ανέλαβε και τις έφερε όλες εις πέρα θετικά. Πολλές θετικές ε, παρατηρήσεις, σωστή πορεία προς τον εκδημοκρατισμό με κάποια όρια βεβαίως και περιορισμούς όπως αυτά που υπενθυμίστηκαν και τα οποία δεν θα ε, αναπτύξω κι άλλο. Η ψηφοφορία ε, πήγε καλά, έδειξε ότι ο λαός έχει συνέστηση του τι συμβαίνει, καταλαβαίνει τι διακυβεύεται, τι ψηφίζει. Και ήθελε να είναι πρωταγωνιστής αυτής της ιστορικής μετάβασης για την Βυρμανία, που νομίζω ότι είναι και αμετάκλητη. Απλώς να πω και το εξής. Προσοχή και πάλι προσοχή και άλλη προσοχή. Διότι είναι αμετάκλητη αυτή η πορεία, αλλά είναι μια πορεία μετάβασης. Και εδώ χρειαζόμαστε και υποστήριξη με όλη την απαραίτητη εξισορρόπηση των διαφορετικών τάσεων. Διότι πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκινάει από χαμηλά με τους αγώνες του λαού, ε, με την ε, Ανσουσί, Σούγη, ε, με τους αντιφρονούντες που φυλακίστηκαν και όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα. Η στρατηγική της πορείας αυτής επιβεβαιώθηκε και ε, εκφράστηκε και από τους στρατιωτικούς με μια κυβέρνηση που για πρώτη φορά είχε και πολιτικό χαρακτήρα, εκπροσωπούσε την, πολιτεία, την κοινωνία των πολιτών. Μια πρώτη, ένα πρώτο ρεκόρ για την ε, Μιανμάρ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται το σωστό σημείο ισορροπίας, διότι μπορεί να υπάρξουν και ε, αντιδράσεις από την πλευρά των στρατιωτικών που για την ώρα διατηρούν την εξουσία τους. Τα προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώτε λοιπόν είναι η μεταρρύθμιση του συντάγματο και θα κλείσω αυτά. Ε, με, τροποποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω μιας πολιτικής συμφωνίας που είναι απαραίτητη και αναγκαία. Διότι, όπω είπα, υπάρχει ακόμη το δικαίωμα ανησυχία από τους κριτικού. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Όπως υπόθηκε, το κόμμα του LND που κέρδισε. Ε, δεν έχει ακόμα λύσει όλα τα προβλήματα. Συναντήσαμε έναν δημοκράτη στρατηγό, μια εξέχουσα προσωπικότητα της χώρας σύμβολο, ε, πραγματικό, αλλά πέραν αυτής της δημοκρατικής πραγματικότητας δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει μια χειροπιαστή έκφραση του τι σκοπεύουν να κάνουν, διότι οι επενδύσεις φτάνουν στη Γερμανία και είναι επενδύσεις που έχουν έρθει από ε, ψηλά ε, που στις περιφέρειες και τις επαρχίες πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα στους κατοίκους και τον πληθυσμό. Το πρόβλημα επίση, τα προβλήματα παραμένουν ε, τα θέματα του πολέμου, τη ενόπλης σύραξη. Υπάρχει πόλεμο στην Μιανμάρ, ακόμη υπάρχει πόλεμο πόλεμος, εθνοτικές ε, μειονότητε που ε, έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις, 10.000 μαχητέ, διαφορετικών εθνοτικών, εθνοτικών μειοτήτων σε σχέση με τι 60.000 που υπάρχουν. Ξέρουμε τι γίνεται στα κρατήρια του Βορρά, στο Σαν και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων. Θα πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή κοινότητα να αναλάβει την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Να δούμε τι γίνεται και στα σύνορα Ταϊλάνδης και Γερμανίας. Ε, μιλάμε για ανθρώπους χωρίς κανένα μέλλον, διότι δεν τους αναγνωρίζεται το καθεστώς τους ούτε στην Ταϊλάνδη ούτε στην Γερμανία. Βρίσκονται λοιπόν σε ένα ε, απόλυτο μηδέν και να ζουν στο κενό. Ε, αυτό είναι ένα πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα Γκόμες. Μεγάλο σεβασμό έχω για την ομάδα της, την διακομματική που συμμετείχε ως ε, παρατηρητές στις εκλογές, κάτι που είναι εξωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των εκλογών. Πραγματικά οι σχέσεις μας ε, με αυτήν τη χώρα λόγω της ρητορικής μίσους, της ε, θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας, της στρατιωτικής δικτατορίας, του ζητήματος των Χίνγκια. Εγώ δυστυχώς εξαιτία όλων αυτών των καταστάσεων δεν είμαι ιδιαίτερα ε, αισιόδοξο ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση για τις μειονότητες. Παρά την πλειοψηφία του NLD στο Κοινοβούλιο, ε, ένα ζήτημα που θα ήθελα να, ρωτήσω την Άννα είναι το εξή. Θυμάμαι ότι η Αν Σανξουξή δεν επετράπει να ε, ε υποψηφιότητα για πρόεδρος ε, λόγω του ότι τα παιδιά της έχουν βρετανική υποψηφιο, υπηκότητα. Ποιες είναι οι δυνατότητες, πιθανότητες να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Θα ασκήσει την εξουσία της μέσω αντιπροσώπου ή θα υπάρξει δυνατότητα να ε, αναθεωρηθεί το Σύνταγμα προκειμένου να μπορεί κάποια στιγμή να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Παρακαλώ έχει καταθέσει ο καλεσμένος μας. Γι' αυτό οι υπόλοιποι χρόνου φίδου. Ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ. Θα είμαι επιγραμματικός. Είναι σαφές ότι η προσέλευση στις κάλπες ήταν ικανοποιητική, συμμετοχή των γυναικών επίσης, η συνεισφορά τους μεγάλη. Το πρόβλημα είναι οι μειονότητες, η συμμετοχή τους. Η Ροίγκα, για παράδειγμα, η μουσουλμανική κοινότητα. Ε, μέχρι και κατηγορίες για γενοκτονία έχουν ε, αναφερθεί. Και παρόλα αυτά η, η διεθνής κοινότητα σιωπεί. Οπότε πού στηρίζετε την ε, ελπίδα σας ότι με τις εκλογές και το αποτέλεσμα θα αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. είναι απαράδεκτο ο στρατός να έχει 25% των εδρών του Κοινοβουλίου και δικαίωμα άρνηση κυρίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για να Γκόμες, αλλά παρακαλώ λακωνικότατα. Θα ήθελα να απαντήσω στον Τσάρλ Τάνοκ. Όπως είπε και ο, Λα, ο, ο κύριος Λάμστορφ, αυτό είναι ένα αντιδημοκρατικό και προτάκουστο χαρακτηριστικό του συντάγματος, αλλά και άλλα σημεία του συντάγματος χρήζουν αναθεώρηση. Το 25% των εδρών για το στρατιωτικούς, η παρουσία τους ε, στην κυβέρνηση, το ΒΕΤΟ. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρόκληση του κόμματος NLD να επανέλθει στη δημοκρατική διαδικασία και φυσικά θα πρέπει να αποκτήσει και τις ε, δεξιότητες για την άσκηση της εξουσίας, γιατί και στη διάρθρωση του έχει πολλές δυσκολίες. Γιατί η Αγκ έχει κορυφαίους συμβούλους, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει το κόμμα της να έχει καλύτερη δομή, κάτι που δεν ε, το έχει εξασφαλίσει ακόμη κύριος Λάμστορφ. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία για τα επίμαχα σημεία και τα τροτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για την πολύ καλή συνεργασία και να τονίσω την ανάγκη ε, παρακολούθησης της ε, δημοκρατικής διαδικασίας. Το Κοινοβούλιο θα το κάνει μέσω της κυρίας Σαρχεντίνη. Και χθες στην ομιλία που έκανα ε, θα είναι τα κρατημέλη να κάνουν το ίδιο για να στηρίξουμε τη χώρα στην προσπάθειά της. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο που προβλέπει η ανταλλαγή απόψεων με τον Γιασίν Μπραχήμ που είναι Υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας ε, Ανάπτυξη και Επενδύσεων στην Τινησία. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την ευκαιρία αυτή για ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς άλλωστε το ζητήσατε για να μας παρουσιάσετε το στρατηγικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων για, το 2000, για την περίοδο 2016-2020. Επίσης θέλαμε να σας εκφράσουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας για προς τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων που έγιναν στην Τίνιδα στις 24 Νοεμβρίου. Που δυστυχώς ήταν η τρίτη φέτος τρομοκρατική επίθεση. Θα ήθελα να πω ότι συμμετέχουν εδώ και τέσσερα μέλη της Τινησιακής Βουλής με αντιπροσωπεία και μέλη της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός υπέστη πλήγμα μετά από τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, χάνοντας έτσι ένα σημαντικό οικονομικό εισόδημα. Και μάλιστα υπήρχαν προβλήματα και με τις ε, εξαγωγές. Ε, κλονίστηκαν βασικές ε, αξίες όπως η ανεξιθρησκεία, η ανοχή, ε, προστασία των γυναικών, των παιδιών. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο μιας δημοκρατίας και η αποκέντρωση των εξουσιών είναι σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας. Επίσης, Χρειάζεται διαφοροποίηση της οικονομίας, πρόθεση του επιχειρηματικού πνεύματος, αύξηση των εξαγωγών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίου και εξάλληψη των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της Τινησίας, ιδιαίτερα μεταξύ των παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας. Χρειάζεται επίσης μια χρηστή και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και ευπρόσδεκτα και από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ε, μέσα και χρειάζονται για τη χρηματο, μακρο, μακροχρηματοπιστωτική στήριξη της χώρας. Περιμένουμε λοιπόν την παρουσίαση των ε, μεταρρυθμίσεων και να σας διαβεβαιώσω για την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τη χώρα σας και στην προσπάθειά σας να εδραιώσετε τη δημοκρατική διαδικασία. Μάλιστα, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ε, θα μεταβεί στην Τινησία στις 6 και 7 Ιανουαρίου. Αυτά. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Ένα δεκάλεπτο σας αρκεί, το θεωρείτε αρκετά γενναιόδωρο. Ευχαριστώ πολύ. Μου δώσαν τη δυνατότητα να μιλήσω ε, όποια γλώσσα θέλω και μιας και έχετε τη δυνατότητα θα μιλήσω γαλλικά αν μου το επιτρέπετε. Χαίρετε, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη χώρα μας, την Ισία. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι στις 17 Φεβρουαρίου 2011, τρεις μέρες μετά την ε, ε, φυγή του Προέδρου οργανώσατε και αφιερώσατε την Ολομέλεια, τη Σύνοδο του Θεσμικού σα στην Τινησία. Χαιρετήσατε τότε τον, το, την τόλμη του λαού της Τινησίας και εκφράσατε την προθυμία του Ευρωκοινοβουλίου να βοηθήσει την Τινησία στην δημοκρατική τη πορεία. Και αυτό όχι μόνο το πράξατε, αλλά με πολλέ επιτόπου επισκέψει στην Τινησία κατά τη φάση τη δημοκρατική μετάβαση για να δείτε, να παρακολουθήσετε τι συμβαίνει στις εκλογές με μέλη της κυβέρνησης και την ίσιους βουλευτές κάποιοι βρίσκονται σήμερα μαζί μας και τις συνομιλίες επαφέ που είχατε μαζί τους δείχνετε την προθυμία να μας στηρίξετε. Η Ευρώπη στην ιστορία της, την πρώτη σφατή ιστορία τη, έζησε την δημοκρατική μετάβαση πολλών χωρών, οπότε γνωρίζει ότι δεν είναι ποτέ απλέ και εύκολες. Πού έχουμε φτάσει λοιπόν στην Ισία. Στην ε, πρώτη περίοδο με την ε, ε, συνέλευση την συνταγματική καταλήξαμε να εγκρίνουμε το 2014 το σύνταγμα και με μία ε, συνέλευση, εθνοσυνέλευση για πέντε χρόνια, καθώς και έναν ε, πρόεδρο για πέντε, για πέντε ετή θητεία. Έτσι φτάσαμε ένα πρώτο στάδιο της θεσμικής ε, πρόοδου. Μπορέσαμε λοιπόν να βρούμε μία σχετική ισορροπία. Μία ισορροπία όπου όλοι στην κοινωνία συμφωνούν να συμβιώσουν, αλλά βεβαίως όποτε υπάρχει μια συνελευση εθνοσυνελευση για πεντε χρονια καθως και εναν προεδρο για πεντε για πεντε ετσι φτασαμε ενα πρωτο σταδιο της θεσμικης προοδου ξανααναδύονται οι διαφωνίες. Αυτή τη στιγμή το στοιχείο της ασφάλειας και οι επιθέσεις που ζήσαμε φέτος είναι στοιχεία που όξυναν τις ε, διάφορες διελκυστίνδες που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πάντως για την καλοσύνη σας. Δυστυχώς και εγώ θα πρέπει εξ ονόματος της τη ελληνική κυβέρνηση να σα εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για όσα συνέβησαν στην Ευρώπη, ιδίω στο Παρίσι. Συγγνώμη, και αν δούμε τι συνέβη του τελευταίου τρεις μήνες στο Λίβανο, στην Τουρκία ή στην Τινησία, Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κίνδυνο, μια πρόκληση πολύ σοβαρή, η οποία ονομάζεται τρομοκρατία. Και θα πρέπει από κοινού να την πολεμήσουμε. τα τελευταία πέντε χρόνια που φτάσαμε, ελευθερία έκφρασης. Ε, κάποιοι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ των ε, καλύτερων. Ε, και σε κάποιες υπερβολές που τις δεχόμαστε και τις ε, αποδεχόμαστε. Βεβαίω, θα πρέπει τώρα να πάμε πιο ε, μακριά, πιο πέρα. Η κοινωνία μας αρχίζει να εκφράζει ανυπομονησία σε σχέση με τι κοινωνικέ και οικονομικέ τη μέρημνε. Γι' αυτό η κυβέρνησή μα επέλεξε να προχωρήσει και να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερω στο πρόγραμμα για την ερχόμενη πενταετία, ε, το οποίο θέλουμε να εντοπιστεί στο σωστό πλαίσιο. Ξεκινήσαμε με αυτό που ε, ονομάστηκε σημείωμα προσανατολισμού, το οποίο θα σας παρουσιάσω σύντομα και αυτούς τους προσανατολισμούς τους έχουμε αναπτύξει σε ένα στρατηγικό λεπτομερές πρόγραμμα με το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται, το σύνολο των διατάξεων και των στόχων καθώς και μια σειρά από στρατηγικά προγράμματα για την περίοδο 2016-2020. Το πρόγραμμα αυτό θα περάσει από την κυβέρνηση θα φύγει από την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο τον Μάρτιο και Απρίλιο. Ελπίζουμε ότι μετά με μια διεθνή διάσκεψη στις 2 και 3 Ιουνίου του χρόνου θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το πρόγραμμα αυτό και να έχουμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας ώστε να έχουμε και τα μέσα να εκτελέσουμε σωστά το πρόγραμμα αυτό. Εάν λοιπόν μου επιτρέπετε θα περάσω απευθεία την διαφάνεια παριθμών 6 για να κερδίσουμε χρόνο, επειδή δεν έχουμε και πολύ, και θα ξεκινήσουμε από την διάγνωση, αυτή που ε, αναφέρεται στη διαφάνεια 5. Στην προηγούμενη, ε, όχι σε αυτή. Η διάγνωσή μας λοιπόν θα καλύπτει όλη την περίοδο ανάπτυξη της Τινησίας. Η Τινησία είχε ανάπτυξη 4% μέχρι το 1984 και του 2010. 4% ε, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Ε, είναι υψηλό φαίνεται αυτό το ποσοστό και έτσι είναι. Αυτή η ανάπτυξη όμως δεν ήταν ε, σωστά κατανεμημένη. Η, το ποσοστό αυτό και στην Τινησία ήταν 2% την ίδια περίοδο και γι' αυτό στο τέλο τη Επανάσταση είχαμε όχι απλώ ένα μεγάλο ποσοστό ανεργία αλλά και μια χώρα διχασμένη. Ο Βορρά και η Ανατολή ήταν ε, σε σχετικά ανεπτυγμένοι ενώ τα Δυτικά και ο Νότο ε, πολύ λιγότερο ανεπτυγμένοι. Ε, γι' αυτό ξεκίνησε από το κέντρο και τα κέντρο-δυτικά η Επανάσταση. Η μη συμμετοχική αυτή ανάπτυξη μα κόστησε πολύ ακριβά. Ε, Επίση, επιτείνεται από ένα ποσοστό ανεργία των πτυχιούχων τη ε, ανώτατη εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι κάπω έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό μα σύστημα, για να το πούμε έτσι. 30% έχουμε φτάσει φέτο με το ποσοστό ανεργία των ε, πτυχιούχων επενδύσεις. Ε, το κράτος επένδυσε 8% του ΑΕΠ, επενδύσει, επενδύσεις, μέχρι το 2000 και μετά έγιναν ε, επιλογές να μειωθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Ο Μπεναλή ε, έκανε πολλές κακές επιλογές, αλλά τουλάχιστον δεν άφησε κακά δημοσιονομικά. Μόνο 35% χρέος ε, ως προς το ΑΕΠ και με μη κρατικέ επενδύσεις, ώστε οι περιοχές δυτικά και νότια να φτάσουν το επίπεδο ανάπτυξης του ε, της Ανατολής και του Βορρά της χώρας, των παράκτιων περιοχών. Μετά την Επανάσταση λοιπόν οι επενδύσεις ήταν ασταθείς, οι ιδιωτικές ιδίως ε, ε κάμφθηκαν. Ε, για να σας δώσω μια ιδέα, δημόσιες επενδύσεις παρουσιάζουν 40% ακόμη, πολύ σημαντικό ποσοστό, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις από την Τινησία φτάνουν το 45% Τη 115% έμεσα ξένε επενδύσει. Πολύ χαμηλό ποσοστό, κυρίω για την ενέργεια. Ω προ την περιφερειακή ανάπτυξη, δυστυχώ δεν υπάρχει η σωστή συμπερίληψη. Το βλέπετε και σε αυτό το χάρτη. Βλέπετε ότι τα ανατολικά και ο τη χώρα είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι από ότι τα παράκτια, τα παράλια. Ε, το θεσμικό πλαίσιο ε, οδήγησε σε αύξηση του παράλληλου εμπορίου στη χώρα μας, μια αύξηση της πλουτοκρατίας όπως ονομάζεται και του νεποτισμού, αλλά και η αποδυνάμωση των ε, θεσμών πριν την Επανάσταση οδήγησαν σε περισσότερη διαφορά. Αυτό είναι μια πρόκληση για το μέλλον. Η κοινωνική μας πολιτική είναι αρκετά παρεμβατική, με την έννοια ότι υπάρχει στήριξη λόγω της ε, ισχυρής παρουσίας της μεσαίας τάξης και αυτό είναι μια επιλογή που έγινε με την ανεξαρτησία τη ε, Τινησία. Αυτή η μεσαία τάξη εντωμεταξύ όμω έχει φτωχύνει τα τελευταία χρόνια παρά το 20% του ΑΕΠ σε κοινωνικά επιδόματα. Αυτό θα πει ότι ε, τα δημόσια προγράμματα κοινωνική κατανομή του πλούτου ε, ε, ε πετυχαίνουν εν το στόχο του. Έχουν πληγεί πολλά στρώματα τη κοινωνία βέβαια τα τελευταία πέντε χρόνια γιατί κάναμε την επιλογή ασχέτω κυβέρνηση μια υποχρεωτική επιλογή, και αυτό προέκυψε λόγω της επανάστασης και των κοινωνικών ανισοτήτων που εντόπισε, κοινωνικές ανισότητες οι οποίες ήταν συστηματικές ω προς τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων κλπ, αλλά και το γεγονός ότι η λίγη ανάπτυξη που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή το 5% ε, κατά μέσο ε, ήταν κάτι που το στήριξε η κατανάλωση, διότι οι επενδύσεις ε, μειώθηκαν πολύ και το ίδιο και οι δαπάνε του κράτους. Ως προς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο ζήσαμε, είδαμε ότι υπήρχε μεγάλο προσανατολισμό όλων των επενδύσεων προ τα παράκτια, τα παράλληλα τη χώρα, αλλά εκεί ε, υπήρξε μια διόγκωση των αστικών κέντρων με επενδύσεις όπως η χημική βιομηχανία, η, η περιοχή του ΣΠΑΚΣ και του ΚΕΜ, οι οποίες στηρίχθηκαν ιδιαίτερα από αυτή τη βιομηχανία όπως και τις χάφησα στα εσωτερικά της χώρας και υπήρξε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών της χώρας το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η Τινησία όπως τα ξέρετε έχει πολύ ισχυρού δεσμού με την Ευρώπη. Η οικονομία μα όμω από τη συμφωνία που υπογράψαμε μαζί το 1996 και η οποία μα έδωσε μεγάλη όθηση τελικά δεν υπήρξε σωστή διαφοροποίηση ω προ το άνοιγμα των αγορών. Παρά ε, τι κινήσει τη Ευρώπη η Τινησία παρέμενε αρκετά συγκεντρωμένη με 70% των συναλλαγών τη να επικεντρώνεται σε τέσσερι ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, σε δύο διαφάνειε παραπέρα βλέπουμε τα εξή. Στο μέλλον θα ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την οικοδόμηση της χώρας όπως την έχουμε αντιληφθεί. Οι θεσμοί μας ακόμη ε, βρίσκονται σε φάση οικοδόμησης. Το Κοινοβούλιο μόλις ψήφισε τις τελευταίες εβδομάδες το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και το Συνταγματικό Δικαστήριο. Είναι σημαντικό αυτό για την τρίτη εξουσία να αρχίσει να αναλαμβάνει καθήκοντα και έχουμε και άλλους σημαντικούς θεσμούς όπως ε, το όργανο για την καταπολέμηση της διαφθοράς η, η ασφάλεια για τις επόμενες γενιές, θεσμικά όργανα, θεσμοθετημένα που θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται τα ερχόμενα χρόνια. Επίση, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει κοινωνική σταθερότητα και ένα κλίμα για να μπορούν οι φορεί και οι θεσμοί να ε, διοργανώνουν κοινωνικό διάλογο. Δυστυχώ, ακόμη έχουμε αντιπαράθεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των ε, ίδιων των εργοδοτών με την κυβέρνηση. Παρά το γεγονό δηλαδή ότι οι εταίροι αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιό μας και είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για τον ε, διάλογο αυτό τον οποίο καταφέραμε να έχουμε για να μπορούν οι πολιτικοί ευθύνοντες να μιλούν μεταξύ τους αλλά σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο ε, στο επίπεδο των επιχειρήσεων έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε τα ερχόμενα χρόνια. Επίσης, Έχουμε να καθορίσουμε συγκεκριμένε επιλογέ για, ε, για του στρατηγικού προσανατολισμού του κράτου. Ο ιδιωτικό τομέα έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει ω κριτήρια δύναμη τη ανάπτυξη και πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη, όπω ήδη συμβαίνει στην κοινωνική οικονομία στην χώρα μα. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να διδραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο τα ερχόμενα χρόνια. Τώρα θα περάσω απευθεία στη διαφάνεια 13-14 για να μιλήσω για του άξονε ανάπτυξη για το μέλλον. Την προηγούμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη δική μας θεώρηση για το μέλλον, ε, στο επίπεδο της κυβέρνησης και με διακομματική στήριξη, τον συνασπισμό που αυτή τη στιγμή κυβερνά. Δηλαδή έχουμε πέντε άξονε μπροστά μα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην καλή διακυβέρνηση, τη χρηστή διακυβέρνηση και τι φιλόδοξε μεταρρυθμίσει που ήδη έχουν ξεκινήσει από δύο-τρία χρόνια και πρέπει να επιταχυνθούν. Βλέπουμε, πάμε στην επόμενη διαφάνεια, δύο διαφάνειε παραπέρα, 15, ε, ακόμη πιο πέρα, ευχαριστώ. Ε, βλέπουμε ότι χρειάζεται να γίνει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων, κυρίω οικονομικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξοικειωθούν οι κρατικέ τράπεζε. Ε, θα πρέπει να περάσει σύντομα από το Κοινοβούλιο ένα νέο νόμο για τι τράπεζε. Έχουμε φορολογική μεταρρύθμιση η οποία ξεκίνησε από 2-3 χρόνια και κάθε φορά που υποβάλλεται ένα σχέδιο προπολογισμού ε, γίνονται βήματα προόδου για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση των ε, τελωνίων για να καταπολεμήσουμε την παράλληλη την κρίζα αγορά. Θα πρέπει το τελεινικό μα σύστημα, οι φορολογικοί δασμοί να αναθεωρηθούν ώστε να πλήξουμε την παράλληλη αγορά, όχι μόνο όμω τιμωρητικά, αλλά και με θετικά κίνητρα, ε, βελτιώνοντα του τελικού μα δεσμού. Ο κώδικα των επενδύσεων, είναι, ο νόμο για τι επενδύσει θα περάσει από το Κοινοβούλιο, θα συζητηθεί σύντομα και θα πλουστευθούν, θα διευκρινιστούν καλύτερα οι κανόνε πρόσβαση στην αγορά μα. Θα υπάρχει ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την προάσπιση των επενδυτών και για να μπορούν να έχουν απλούστερε διοικητικέ διαδικασίε μπροστά του. Με τα απαραίτητα οικονομικά εργαλεία για να ενθαρρυνθούν και ιδιωτικέ μεταρρυθμίσει χρειάζονται και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να γίνει η σωστή διασύνδεση μεταξύ τη εκπαίδευση, τη επαγγελματική κατάρτιση και του πανεπιστημιακού συστήματο. Έχουμε σοβαρή υποχώρηση τα τελευταία 15 χρόνια σε αυτό το σκέλο. Θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα στήριξη που μα έδωσε εδώ για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μα συστήματο. Το υγειονομικό. Και αυτό ω προ την αποτελεσματικότητα και ω προ τι επιτυχίε. Έχουν προβλεφθεί μια σειρά από μεταρρυθμίσει που θα επιταχυνθούν την ερχόμενη πενταετία. Υπάρχει λοιπόν ένα εργοτάξιο, θα έλεγα, μπροστά μα, πολύ ευρύ και ο κάθε τομέα, ο κάθε κλάδο θα έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μεταρρύθμιση του και με τα πάρετε εργαλεία για να υποστηριχθεί αυτό. Η ίδια κυβέρνηση περνάει βεβαίω και από τη διαφάνεια και το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών για να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν και τι εξελίξει. Αυτό θα το δούμε στι δημοτικέ, περιφερειακέ και τοπικέ εκλογέ. Χρειάζεται από συγκέντρωση για να υπάρχει μεγαλύτερη εγκύτητα των πολιτών με την εξουσία, με τους πολιτικούς ευθύνοντες. Την επόμενη διαφάνεια οικονομία. Η οικονομία της Τινησίας θεωρείται χαμηλού κόστους, με λιγότερο ακριβέ συνθήκες διαβίωση, χαμηλούς μισθούς. Θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτή την εικόνα και να εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε ένα hub οικονομικό, ένας κόμβος. Ξεκινά να γίνεται αυτό, ιδίω στην αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε από τις χώρες, από τις πιο σημαντικές χώρε που εξάγουν αυτοκίνητα. Σε ορισμένου κλάδου, σε ορισμένες αγορές ε, ε, πολύ εξειδικευμένε. Το ίδιο και στην αεροναυπηγική. Αρχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερα διπλώματα ευαισθητεχνία στην φαρμακοβιομηχανία. Επίση, σε διάφορε θηγατρικέ έχουμε και εκεί μια ιδιαίτερη θέση και στι τεχνολογικέ υπηρεσίε, είτε για τα λογισμικά, είτε στι εταιρείε των Business Process Operations, είμαστε από του πρώτου έχουμε μια σημαντική ε, γεωγραφική εγκύτητα με τη δική σας αγορά την ευρωπαϊκή, οπότε ε, μπορούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα και με την ε, ενδυνάμει αφρικανική αγορά με τα εργαλεία που διαθέτουμε στην Τινησία. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε ένα hub, ένα κομπικό σημείο για τι εμπορικέ συναλλαγέ, ε, ξεπερνώντα τι καθυστερήσει που είχαμε ω τώρα στην διοργάνωση κυρίω, τη λογιστική. Ε, οι εταιρικέ σχέσει δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο, αλλά είναι μόνο δημόσιε. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε προ την ανάπτυξη. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε προ την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συμπερίληψη. Σήμερα, όπω τα ξέρετε, η Τινησία έχει ήδη πραγματοποιήσει πολύ μεγάλο έργο ε, για τα δικαιώματα των γυναικών που προστατεύονται. 28% ε, ε, σήμερα των εργαζομένων στην Τινησία είναι γυναίκες. Είναι χαμηλό το ποσοστό, αλλά από αυτό το 28% θέλουμε να περάσουμε στο 35% στο 2020. Υπάρχει αγύραση του πληθυσμού. Είναι ο μέσος όρος ηλικία 31 ετών στην Τινησία σήμερα. Οι γυναίκες μπορούν να μα βοηθήσουν να πετύχουμε καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων και να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση κυριαρχίας του πληθυσμού μα. Η τιμήση στο εξωτερικό έχουμε και εκεί πολλά προγράμματα φιλόδοξα, διότι αυτή τη στιγμή, όπω είπατε, υπάρχει πτώση στι τουριστικέ δραστηριότητε. Η πρώτη πηγή ξένου νομίσματο για την Τινησία είναι τα εμβάσματα των Τινήσιων μεταναστών, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πρέσβει μα και είναι μία δύναμη που μας επιτρέπει να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στις χώρες όπου κατοικούν εκείνοι. Η πολιτιστική διάσταση, ο πολιτισμός αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά παρόν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θέλουμε και αυτή η διάσταση να ενισχυθεί και να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην ιστορία της Τινησίας. Την ιστορία της ανθρωπότητας τη διδασκόμαστε στην Τινησία, διότι είναι χιλιετή η ιστορία της χώρας μας και αυτό έχει αξιοποιήσει και ο ταινισιακός τουρισμός για να ε, παρουσιάσει μεγαλύτερη προσφορά με την ιστορία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Τινησίας. Έχουμε λοιπόν φιλόδοξα προγράμματα για την αγωγή επίσης του πολίτη και με προγράμματα αθλητικά και πολιτιστικά. Και ο κοινωνικός διάλογος είναι για μας μια πραγματική πρόκληση. Η Ευρώπη μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ εδώ. Θέλουμε μια άλλη φιλοσοφία κοινωνικού διαλόγου, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που συνήθως συμβαίνει μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών είναι μια διελκυστή δυνάμεων. Θέλουμε να περάσουμε σε μια νέα νοοτροπία λοιπόν. Μια νοοτροπία συμμετοχική των εργαζομένων στο σύστημα, το οικονομικό σύστημα υπό την ευρία έννοια. Δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε τους άλλους δύο άξονες, εάν μπορούμε να πάμε στη διαφάνεια για τις ε, επαρχίες, τις περιφερειές, βλέπουμε ότι το κράτος ε, επενδύει σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο έργων, ηλεκτρισμός, ίδρευση, ε, εκπαίδευση, υγειονομικά για όλον τον πληθυσμό. Όμω οι ιδιωτικέ επενδύσει δεν βρίσκονται στη ίδιο ύψο. Γιατί βλέπουμε μετά από μελέτε και τα διάφορα πορίσματα που έχουμε ότι δεν υπήρχαν αρκετέ υποδομέ που να επιτρέπουν τη διασύνδεση των ε, επαρχιών με τα παράλια. Είμαστε μια μικρή χώρα, ό,τι παράγουμε πρέπει να εξάγεται ώστε ο επενδυτή να έχει κίνητρα να πάει να παράγει στι διάφορε επαρχίε και να μπορεί να φτάσει και στα λιμάνια πολύ εύκολα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη ακτή, 250 χιλιόμετρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, ε, το πιο ε, μακρύ. Ε, εδώ λοιπόν είτε οι σιδηρόδρομοι είτε οι οδικές διασυνδέσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το δίκτυο που θα συνδέει τον Νότο με τα παράλια της χώρας. Και τέλος, όχι το πιο σημαντικό αναγκαστικά, γιατί δεν τα έχω βάλει με ιεραρχική σειρά, η ε, πράσινη οικονομία θα είναι ένας πυλώνας της ανάπτυξης για το στρατηγικό μας πρόγραμμα στο μέλλον. Ξέρετε ότι την Ισία είναι μια χώρα άγωνη, δεν έχουμε υδάτινους πόρους και έχουμε πολλές δυσκολίες ε, θέλουμε στον άξονα αυτό να δώσουμε έμφαση στα εργοστάσια, εργοστάσια αφαλάτωσης στα παράλια, διότι εκεί είναι πιο λογικό, θα ε, βελτιστοποιήσουμε την διαχείριση των ε, υδάτινων πόρων μας και κυρίως να φέρουμε νερό από το βορρά προς τα νότια της χώρας. Ε, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαχείριση εκεί. Στην ενέργεια έχουμε καθυστερήσει σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Παράγουμε μόνο 3% του ηλεκτρισμού μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε στο 2020 να φτάσουμε το 12% και θα φροντίσουμε να περάσει νομοσχέδιο από το Κοινοβούλιο με ένα προεδρικό διάταγμα εκτέλεσης. Έχουμε εργαστεί πολύ σε επίπεδο εταιρικών σχέσεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Έχουμε καθυστερήσει και με τη βιομάζα και την διαχείριση αποβλήτων, αλλά θα εκμεταλλευτούμε για τις δημοστικέ αρχές αυτή τη στιγμή το φιλόδοξο πρόγραμμά μας για να έχουμε μια καλύτερη αποκομιδή και ανακύκλωση διαχείριση των αποβλήτων. Το ίδιο και για τους υδατινούς πόρους. Πολύ πίεση υπάρχει στα παράλια με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την ε, ερημοποίηση στα νότια της χώρας. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με το πρόγραμμά μας και για να προστατευτούμε από αυτά τα ε, περιβαλλοντικά φαινόμενα. Ε, η τελευταία διαφάνεια, το πρόγραμμα ανάπτυξη για το 2016-2020. Βεβαίω είμαστε εκτεθειμένοι, βεβαίω υπάρχουν παράγοντε κινδύνου, όμω κάναμε την επιλογή στο επίπεδο τη στρατηγική μα θεώρηση να είμαστε ρεαλιστέ και πραγματιστέ. Να έχουμε ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, την, το καλύτερο σενάριο για να το πω έτσι. Ένα πρόγραμμα ανάκαμψη μέσω των επενδύσεων, μέσω στο προγραμματισμό και εκτέλεση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Ξεκινάμε με ένα ανώφλη το 2016 μεταξύ 0,25% ανάπτυξης και με ε, όσα συνέβησαν φέτος λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Είναι φιλόδοξη αρχή για το 2016. Το 2017 θα έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό και επιτάχυνση από το 2018. Το πρόγραμμα αυτό βεβαίως θα λάβει σαρκακοστά μόνο εφόσον φτάσουν οι επενδύσεις που θα πρέπει να τις κινητοποιήσουν αρχικά οι δημόσιες κρατικές επενδύσεις αλλά ελπίζουμε να φτάσουν και οι ιδιωτικές. Είναι θετικές οι προβλέψεις μας διότι απελευθερώσαμε ήδη τον τομέα της ε, διανομής Έχουμε περισσότερο ανταγωνιστικού όρους λοιπόν, θα μειωθούν οι τιμές και για, τη, για τους πολίτες μας και θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Στο επίπεδο του προγράμματος έχουμε προβλέψει δύο σενάρια, αυτό που έχουμε ονομάσει best case, την καλύτερη δυνατή περίπτωση, λαμβάνοντα υπόψη και του παράγοντε κινδύνου και τι δυνατότητε χρηματοδότηση αυτού του προγράμματο, διότι δεν είναι και η πόρη μας. Και ε, αν έχουμε ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα, αν έχουμε τι δυνατότητε να το πραγματοποιήσουμε, μπορούμε να ε, φτάσουμε στην πραγματικότητα σε μια ε, υλοποίηση τη καλύτερη δυνατή υπόθεση, που ελπίζουμε να είναι και αυτή αρκετά θετική. Ναι, uh, Σα ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Παντσέρη, που είναι ο πρόεδρος αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Μακρέπ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω καν πόσο είναι σημαντικό για μας και πόσο μας ενδιαφέρει βαθιά η δημοκρατική μετάδοση της Τινησίας και να υπάρχει και μια θετική ολοκλήρωση αυτής της πορείας. Τονίζω λοιπόν ότι είμαστε στο πλευρό σας και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την οικονομική χρηματοπιστωτική στήριξη που χρειάζεστε και για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που μπορεί να βρίσκονται σε εξέλιξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτήν την έννοια να πω ότι προσπαθούμε να πείσουμε και τους ευρωβουλευτές και για το θέμα του ελαιόλαδου που για μας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην Τινησία. Πρέπει να γίνουν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επενδύσεις. Διότι κατά την άποψή μας και το έχουμε επαναλάβει ξανά και ξανά ε, με όλα τα περιλήγματα για να το πω έτσι η πραγματικότητα ε, επιβάλλει να συνεργαστούμε με την Τινησία. Δύο παρατηρήσεις εδώ. Φοβούμαστε δύο πράγματα ως προς την οικονομία της Τινησίας και κυρίως των κλάδων υπηρεσιών. Η Αλία, ένα παράδειγμα δίνω, ακόμη δεν είναι ανταγωνιστικός ο τομέας αυτό σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Ε, με τις διαφάνειες που μας παρουσιάσατε είδαμε ότι πραγματικά χρειάζονται οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Εάν πρέπει να αποστείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα, είναι ότι η πορεία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να επιταχυνθεί. Είναι ζωτική σημασία, όχι μόνο για μα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Και δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού συστήματο πρέπει να υπάρχει ένα σχετικό επίπεδο ακρίβεια. Να εντοπίσετε προτεραιότητε, τομεί προτεραιότητα όπου πρέπει να γίνουν οι επενδύσει. Δεν μπορούμε να επενδύουμε έτσι παντού πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση για να υπάρξει και όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάπτυξη της θυμησίας. Τέλος, υπάρχει και το θέμα που θίξατε σε, μια από τις διαφάνειες της αποκέντρωσης. Χρειαζόμαστε και πρέπει να δούμε στην πράξη πώς μπορεί να μεταρρυθμίσετε και τα ε, θεσμικά όργανα τους φορείς που θα επιτρέψουν να υπάρξει ομοιογενής ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας. Διότι αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει την Ισία και που παρεμποδίζει την ανάπτυξη ιδίω τη περιοχή τη Πέθρου. Τελευταία παρατήρηση, όπω ξέρετε, μόλις ε, δημιουργήσαμε την εκτή κοινοβουλευτική συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωση της Ισία. Είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Τέλη Γενάρη θα συναντηθούμε για πρώτη φορά Νομίζω ότι αυτό θα είναι σημαντικό όχι μόνο για τι διπλωματικέ μα σχέσει μεταξύ κοινοβουλίων, αλλά και για να υπάρξει υλοποίηση έργου από τα δύο κοινοβούλια για να σα παρακολουθήσουμε στην διαδικασία μετάβαση και να επαληθεύουμε και το πώ προχωρούν οι μεταρρυθμίσει που πρέπει να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κ. Καστάλτο τώρα, που είναι ο εισηγητή τη ΑΦΕΤ για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ισία στο ίσιο ε, περιφερειακό πλαίσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που και πάλι σας βλέπουμε εδώ Υπουργέ Ιμπραήμ και μπορούμε να σχολιάσουμε το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ένα πρόγραμμα πραγματικά πιστικό, φιλόδοξο και που δίνει πολύ θετικές προοπτικές. Αυτό πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην φανούμε κάτω των προσδοκιών σας. Ε, θα πρέπει όντως να πούμε ότι σημαντική στήριξη παράστηκε, έχει προσφερθεί στη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης και ήδη του χρόνου έχουμε προβλέψει αποστολή παρακολούθησης των εκλογών και για τις ε, δημοτικές σας εκλογές. Μα ενδιαφέρει στην Τινησία να δούμε ότι και οι επαρχίε, οι φτωχότερε περιφέρειες, οι μειονεκτούσε, με περισσότερε δυσκολίε, είναι τελείω σωστά διασυνδεμένες με την υπόλοιπη χώρα και μπορούν να αναπτυχθούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο των τοπικών οικονομιών, το πώ λειτουργούν εκεί οι αρχέ, οπότε πρέπει και εκεί να φανούμε παρόντε και να επιμείνουμε στην διαδικασία συνοδείας της όλης της δημοκρατικής προσπάθειας. Είναι επίσης σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις αυτές που αναφέρθηκαν ε, στο πρόγραμμά σας να γίνουν εγκαίρως. Ο χρονικός παράγοντας αυτή τη στιγμή είναι αποφασιστική σημασία. Η Τινησία είναι και θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα ε, για την Αφρικανική Ήπειρο και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Βέβαια είναι πολλοί παράγοντες ε, που αναφέρατε κι εσείς και που θα τον αναμφιβόλω κάποια πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε. Οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να, οι βουλευτές θα πρέπει να βιαστούν και εκείνοι. Ενεργοποιώντας τους θεσμικούς μηχανισμούς, τους φορείς που μπορούν να τους διευκολύνουν. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Να προσθέσω από πλευρά μα, γιατί αναφέρατε μια σειρά από σημαντικού τομεί τη οικονομία που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, τι υποδομέ από τη μία, την διαφοροποίηση της οικονομίας από την άλλη, συμφωνώ σε αυτά. Να μην πέσουμε στο σφάλμα να επικεντρωθούμε σε έναν μόνο ή δύο κλάδους που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Χρειάζεται αρμονική ανάπτυξη της οικονομίας γιατί αυτό θα την καταρτήσει και ανθεκτική σε σχέση με, τα διάφορα, ε, με τους διάφορους τριγμούς, τα χτυπήματα που μπορεί να δεχτεί με τις ε, διάφορες ε, δικημάνσεις της αγοράς. Γι' αυτό και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα είναι σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή θα προτείνουμε ένα ειδικό ταμείο επενδύσεων το οποίο θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο θα επιτρέπει να υπάρχουν διατομεακά προγράμματα που να αφορούν περισσότερο από, ένας, από έναν κλάδους και να ε, δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση και με την κοινωνία των πολιτών. Να μην υπάρχει δηλαδή μόνο εμπορική ε, επικέντρωση, στόχευση, αλλά και τα δικαιώματα του ανθρώπου και των πολιτών να λαμβάνονται υπόψη. Έχει στατηγική σημασία η Τινησία αυτή τη στιγμή και αυτό ξεπερνά και το θέμα των δημογραφικών της χώρας. Σημειώνω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου φαίνεται να το συνειδητοποιεί αυτό όλο και περισσότερο και υπάρχει και το γεγονός ότι δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ε, το θέμα, αλλά και το τι γίνεται και με την ε, γειτονία μας γενικότερα. Δηλαδή, ε, έχοντα υπόψη ότι από τη δική σα ασφάλεια εξαρτάται και δική μα, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση σε αυτή τη σχέση συνεργασία. Γι' αυτό εκφράζω νομίζω την, το γενικό αίσθημα αυτή τη Επιτροπή. Επιθυμούμε να είμαστε παρόντε, να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στην μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση που θα αρχίσει τα πρώτα της βήματα στις αρχές της επόμενης χρονιάς και ελπίζουμε να ε, δημιουργήσουμε μια σταθερή πολιτική σχέση. Είστε η ελπίδα μας. Θέλουμε έναν εταίρο με συνέπεια που να προβάλλει τις αξίες που ε, προσπίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Και όλα αυτά με αμοιβαιότητα και όχι με ε, διχασμούς μεταξύ των δύο παραλίων, βορρά και νότου της Μεσογείου, που φαίνεται να αντιπαρατίθενται και μέσω των εξτρεμιστικών ε, ε, τοποθετήσεων, των εκφράσεων μίσου, αλλά γι' αυτό θα είμαστε και πρόθυμοι να δεχτούμε τις δικές σας θετικέ προτροπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφίσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ε, κύριε Πρεσβευτά, αξιότιμοι βουλευτέ εκτινησίας. Και εγώ είμαι μέρος αυτή τη μεικτή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ισίας. Και θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου η Τινησία ίσως είναι η μόνη χώρα της νότιας όχθης της Μεσογείου που είναι μια πραγματική γνήσια δημοκρατία μεταξύ των υπόλοιπων χωρών ε, της νότιας όχθης της Μεσογείου μεταξύ των αραβικών κυρίως χωρών. Και από αυτή την άποψη για μα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, για άλλου όμω είναι κακό παράδειγμα. Για το Ισλαμικό κράτο, για παράδειγμα, είναι κακό παράδειγμα η Τινησία, γιατί για το Ισλαμικό κράτο είναι η Τινησία ε, ένα παράδειγμα προς αποφυγή για να αναπτυχθεί σε μια αραβική χώρα, μια πραγματική δημοκρατία. Να αυτό κάνει την Ισία. Και γι' αυτό έχει υποστεί το πλήγμα των ε, διαδοχικών τρομοκρατικών επιθέσεων. Και σίγουρα ε, υπάρχουν δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν αυτά που επιχειρείτε να κάνετε και όλο αυτό το λαμπρό σχέδιο ανάπτυξης που έχετε εκπονήσει για την Τινησία. Το είπατε πολύ εύγλωτα και έχετε βάσιμους λόγους που επιμείνετε σε αυτά τα σχέδια γιατί υπάρχει όντως σημαντική μεσαία τάξη που ναι μεν έχει φτωχύνει αλλά υπάρχει, θα πρέπει να στηριχθεί. Ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ σημαντικός και αυτή η επιθυμία προόδου και προκοπής. Η Τινησία είναι μικρή χώρα, αλλά έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες να πετύχει. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε αφενός τη νέα Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ή ε, συνεργασίας με την Τινησία. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Όπως είπε ο κύριος Καστάλτο, θα πρέπει η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει στην Τινησία, να συμπαρασταθεί στην Τινησία για να στεφθεί με επιτυχία η χώρα αυτή και προσπάθεια της. Ίσως θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα σχέδιο Marshall για να βοηθήσουμε την Τινησία ως Ευρώπη. Και υπάρχει και το θέμα της Λιβύης. Η Τινησία είναι μικρή χώρα και γειτονεύει με μια χώρα που είναι πολύ δύσκολος ε, γείτονας με τεράστια μεταναστευτική ροή που ίσως ε, θέσουν σε κίνδυνο όλα αυτά τα αξιέπαινα σχέδια που μας παρουσιάσατε. Θα ήθελα πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πολιτική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θέλει να σας συμπαρισταθεί, να σταθεί στο πλευρό σας. Το ίδιο και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Βέβαια ε, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Ε, με μεγάλη χαρά σε απευθύνω χαιρετισμό και σε εσά και στα μέλη της αντιπροσωπείας σας και στους βουλευτές. Και πραγματικά το Νόμπελ που πήρε η Τινησία είναι ένα παράδειγμα και επιβράβευση της αιμονής της και της ε, στρατηγικής, ε, του στρατηγικού οράματος που έχει και που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί και να εδραιωθεί η δημοκρατία. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η διάγνωση που κάνατε και το σχέδιο δράση που μας παρουσιάσατε. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Φίσας, η κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα σας είναι πολύ δύσκολη και λόγω της Λιβύης, αλλά όχι μόνο λόγω της Λιβύης. Γιατί η Λιβύη δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό σα, είναι πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω των παραλήψεών τη, λόγω αυτών που αμελήσαμε να κάνουμε μετά την ανατροπή και πτώση του Καντάφη. Η Λιβύη θα είναι πρόβλημα λοιπόν και για μας. Και σίγουρα η Τινησία αυτή τη στιγμή είναι ε, ένα πεδίο δοκιμών για το τι περιμένει την Ευρώπη. Για ένα φαινόμενο που έχει πλήξει με δραματικό τρόπο αυτή τη στιγμή την Τινησία. Αναφερθήκατε στην σημασία που έχει η δέσμευσή σας να εξασφαλίσετε ευκαιρίες για τους νέους, να καταπολεμήσετε τις ανισότητες, να εξασφαλίσετε υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Ε, αναφερθήκατε στους τινήσους μετανάστες, οι περισσότεροι βρίσκονται στην Ευρώπη και όμως αυτή την Ευρώπη που δεν έκανε το καθήκον της, ούτε στη Λιβύη ούτε στη Συρία, επιβάλαμε την πολιτική λιτότητα. Η πολιτική λιτότητα οδηγεί σε φτωχοποίηση, σε αποκλεισμό, σε ανεργία, ιδιαίτερα σε ανεργία των νέων και των νέων την ίσων μεταναστών στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτό έγινε. Φαίνεται ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες ε, στο παιχνίδι που κάνουν και στην... στο αφήγημά τους για τη στρατολόγηση όλο και περισσότερων τζιχαντιστών. Τι, ποια είναι λοιπόν τα λάθη μας που μας εμποδίζουν να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, στην ευημερία και στη μάχη μας υπέρ της νομιμότητας. Ε, όλα αυτά που κάνουμε εμείς επηρεάζουν και εσάς άμεσα και αυτό θα πρέπει να το διατρανώσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σμιθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, Υπουργέ. Βρεθήκαμε ε, στην ε, Τίνιδα μετά την εκλογή σας και χαίρομαι πολύ που βλέπω να προχωράει η κυβέρνησή σας σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές και ξέρετε ότι η Επιτροπή μας ε, υποστηρίζει τις προσπάθειές σας. Με εντυπωσιάζει όμως ότι είμαστε όλοι πολιτικοί και βεβαίως πρέπει να επιστρέφουμε όλοι στις περιφέρειές μας με μια αίσθηση νίκης προόδου ε, εγώ είμαι μέλος ε, και στην ε, Επιτροπή Γεωργίας και είμαι σκιώδης εισηγητής για το ελαιόλαδο και εμείς υποστηρίζουμε τη χώρα σας στον τομέα του ελαιολάδου. Θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν και θέσεις απασχόλησης στον τομέα αυτό. Αλλά πρέπει να κάνετε συγκεκριμένες ενέργειες και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Απολύτως σας έχει υποστηρίξει και οικονομικά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να σας βοηθήσουμε να δείξετε στο λαό σας ότι υπάρχει πραγματική ε, πρόοδος και όφελος από το να ε, ακολουθήσετε τη δημοκρατική οδό. Τι, τι μπορούμε να, εμείς να κάνουμε. Υπήρξε και μια αναφορά στο σχέδιο Μάρσαλ. Εγώ δεν ε, γνωρίζω Εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή πλευρά μπορεί να, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο φιλόδοξη ως προς τη βοήθεια που παρέχει προς εσάς. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κύριε Σεπιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον ε, κύριο Υπουργό και να του απευθύνω μία ερώτηση. Ε, εξοχότατε, ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι ακριβώς η υποστήριξη που έχετε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον ε, τομέα του ελαιολάδου. Έχει ακουστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει πρόταση αυξήσεως της ποσοστώσεως του αδασμολογήτως εισαγωμένου ελαιολάδου από την Τινησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα για τα δύο επόμενα χρόνια προτείνει να εισαχθούν 35.000 τόνοι ελαιολάδου από την Τινησία. Αυτή η εξέλιξη ε, θίγει άμεσα την ε, χώρα μου, την Ελλάδα, η οποία είναι μεγάλη ελαιοπραγωγός ε, χώρα. Και μόνο η ανακοίνωση αυτής της προτάσεως ή αν θέλετε της επιθυμίας για να γίνει αυτή η πρόταση και σε συνδυασμό με την ψυχολογία της αγοράς έριξε κατακόρυφα τις τιμές του ελληνικού ελαιολάδου. Από 4,2 που ήταν μετά 3 3,80 ευρώ τώρα έχει πάει στα 3,20 ευρώ ανά Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άμεσα την οικονομία των 700.000 οικογενειών που ασχολούνται με την παραγωγή του ελαιολάδου στην Ελλάδα και παράλληλα πλήττει και την ελληνική οικονομία, η οποία ήδη βρίσκεται σε ύφεση λόγω των απαραδέκτων μέτρων του μνημονίου που έχει επιβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι δύσκολο σε εμά του Έλληνε να δεχθούμε στα πλαίσια της υποστήριξης μιας εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να γίνουμε συνεργοί σε μια ενέργεια η οποία δημιουργεί συνθήκες αφαιμή του ανταγωνισμού μέσα στην ίδια τη χώρα μας. Θα ήθελα την άποψή σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. And Σας ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω και εγώ από την ε, πλευρά μου εδώ και σας ε, συγχαίρω και για το σχέδιο ανάπτυξης. Πολλοί συνάδελφοι ήδη εξέφρασαν την ε, επιθυμία τους να δουν να, την Τινησία να επιτυγχάνει σε διάφορους τομείς και στις επενδύσεις. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα ε, θέμα. Έχω επισκεφτεί πολλές φορές τη χώρα σας και θα το πράξω και στο μέλλον. Ακούσαμε για την Αραβική Άνοιξη. Αλλά ακούμε και για, την, για τον Αραβικό χειμώνα Φυσικά η χώρα σας κέρδισε το βραβείο Νόμπελ και μου φαίνεται περίεργο το ότι διοργανώθηκαν εκλογές και στη συνέχεια έγιναν δεύτερες εκλογές. Ε, φυσικά σας ε, συγχαίρω για όλα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλοι οι αγώνες που βλέπουμε να διεξάγονται και η συζήτηση για το δημοκρατικό όλαμα στις αραβικές χώρες και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σας ρωτήσω, είναι, είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε την όλη κατάσταση στις και κυβέρνηση, γιατί ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Βλέπουμε όλοι τον, ε, τον, τον πόνο που προκαλεί τον ΤΑΕΣ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά ο μουσουλμανικός κόσμος είναι αυτός που πλήττεται περισσότερο από όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να υπονομεύσουμε το αφήγημά τους και ο καλύτερος τρόπος είναι να αποσαφηνίσουμε ότι η σταθερότητα και η δημοκρατία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι δικτατορίες, η δικτατορία και η αστάθεια είναι από την άλλη πλευρά επίσης όψεις του ίδιου νομίσματος. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να επιτύχετε σε αυτό το δημοκρατικό σας ταξίδι και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο λόγος σας και πάλι κύριε Υπουργέ. Θα είχατε την καλοσύνη να σχολιάσετε ή να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξη που εκδήλωσαν σε αυτή την διαδικασία οικοδόμησης της δημοκρατίας στην Τινησία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε και τη ριζοσπαστικοποίηση, κάτι που θα πρέπει να ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε εκ του ε, τα συμβάντα στην Τινησία, ξέρετε ότι υπάρχει σήμερα ένα πρόβλημα μεταξύ του πληθυσμού για την ε, αξιοπιστία ή την αποδοχή της πολιτικής διαδικασίας και των πολιτικών κομμάτων. Γιατί υπάρχει απογοήτευση. Όταν ξεκινήσαμε ένα διάβημα και ένα χείρημα από, από, τα πάνω, από την κορφή προς τη βάση, δηλαδή συντακτική συνέλευση, ε, σύνταγμα, ε, δημιουργήθηκαν προσδοκίες και μια ανυπομονησία στο κοινό. Και φυσικά στο θέμα της αποκέντρωσης έχουμε παιδίσει πάρα πολλά, γιατί θέλουμε την δημοκρατική μας κουλτούρα να την ριζώσουμε στις περιφέρειες. Γι' αυτό ξεκινούμε από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που ελπίζουμε ότι θα οργανώσουμε το αργότερο στις αρχές του 2017, κατά προτίμηση στα τέλη του 2016. Γιατί η αποκέντρωση είναι πολύ σημαντικό θέμα και αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, γι' αυτό και φαίνεται η άμεση σχέση πολίτη και πολιτική εκεί. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για την αποκέντρωση και συνεχίζεται και η δημόσια συζήτηση και στο Κοινοβούλιο. Βέβαια όλες οι χώρες έχουν περάσει από τα διάφορα αυτά στάδια και είναι μια σταδιακή διαδικασία εγκαθίδρυση της αποκέντρωσης. Έχουμε πάντως μία πρόταση και για τα Δημοτικά Συμβούλια που μάλιστα είχαν εκλεγεί και πριν από την Επανάσταση. Και τώρα θα ξεκινήσουμε ανάποδα, από τη βάση προς την κορύφη. Θα ξεκινήσουμε από τις δημοτικές εκλογές, μετά θα περάσουμε στις περιφερειακές εκλογές και μετά με έμεση ε, ψηφοφορία θα έχουμε 6-7 διαμερίσματα στην Ισία μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων για να ε, αποκαταστήσουμε και να εδραιώσουμε πλήρως τη διαδικασία της αποκέντρωσης. Και προσβλέπουμε στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην προσπάθειά μας αυτή, στο εγχείρημά μας αυτό. Γιατί πολλές χώρες ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία και την έφεραν σε αίσιο πέρας. Ε, η Ιωνή είναι αισιόδοξη και στην Τινησία όσο αφορά την αποκέντρωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αυτή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Ξεκινήσαμε εκ του μηδενός με την πρώτη ε, με την πρώτη συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε την πρώτη συμφωνία του 1996 με την Ευρώπη, που αφορούσε κυρίως τη βιομηχανία και στον απολογισμό που γίνεται ακούγονται και πολλές ε, επικριτικές φωνές, κάτι που δεν είναι δυσάρεστο γιατί το ότι υπάρχουν και επικρίσεις είναι απόδειξη ύπαρξης δημοκρατίας. Πιστεύουμε πάντως ότι με την ε, συμφωνία αυτή θα ενισχυθεί η βιομηχανία της Τινησίας ε, ακριβώς επειδή βρήκαμε συστήματα αντιστάθμισης, μπορούμε να εισάγουμε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μόνο εφόσον ο κατασκευαστής ε, τα μισά αυτοκίνητα που, πολλά, που στην την Ισία τα κατασκευάζει στην την Ισία. Έτσι έχουν έρθει πολλές επιχειρήσεις ε, για να επενδύσουν στην την Ισία, κάτι που θα βοηθήσει την ανάπτυξη και του τοπικού ιδιωτικού κλάδου. Μία ελπίδα που έχει δημιουργηθεί και ελπίζουμε να υλοποιηθεί είναι ότι ε, το ίδιο κάναμε και για τη Γεωργία, έναν κέριο κλάδο της οικονομίας. Βέβαια, την Ισία είναι μικρή χώρα, ένα μικρό τμήμα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Πιστεύουμε όμως ότι με τις συμφωνίες μας θα βρούμε μια κατάσταση αμοιβαίως επωφελή, ώστε να ανοίξουμε τη μικρή την Ισιακή αγορά σε μια αγορά που είναι πολύ πιο μεγάλη ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία και των γεωργικών προϊόντων. Και έρχομαι εδώ στο ερώτημα που θέσατε για το ελαιόλαδο. Σήμερα το ελαιόλαδο, όπως ξέρετε, την νησία για παράδειγμα εξάγει ε, ποσότητες ελαιολάδου μεγάλες προς την Ευρώπη, αλλά και προς ε, Ευρωπαίους εμπόρους ε, που συσκευάζουν και ξαναπολούν το ελαιόλαδο στη διεθνή αγορά. Και διεθνώς η αγορά ελαιολάδου αναπτύσσεται. Και δεν πιστεύουμε ότι η αύξηση των ποσοστώσεων ελαιολάδου ε, της Τινησίας προς την Ευρώπη θα επηρεάσει ιδιαίτερα, γιατί έχουμε ενσωματωθεί ε, αρκετά καλά. Και μάλιστα είχαμε ακριβώς προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή σε μερικές χώρες ε, της Ευρώπης. Γι' αυτό και με ένα προϊόν που έχει συγκεκριμένη αξία και ε, είναι γνωστό σημαντικό ε, και ακριβώς λόγω της άνθησης παγκόσμιας αγοράς δημιουργούνται αμοιβέ ευκαιρίες. Δεν θεωρώ ότι η αύξηση της ε, τινησιακής ποσόστοσης θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δυσμενή αντίκτυπο στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για ελαιόλαδο που το συσκευάσαμε στην Τινησία, που είναι ακόμη μικρότερο ποσοστό των συνολικών εξαγωγών. Και νομίζω ότι δικαιολογείται λόγω της ιδιαιτερότητας η παρουσία του ελαιολάδου στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη και συμπληρωματική προσέγγιση και όχι προσέγγιση με όρους ανταγωνισμού και αντιπαράθεσης. Επίσης, ως προς το θέμα της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, ε, το βλέπουμε ευνοϊκά, γιατί δεν είμαστε μια τόσο σημαντική αγορά που θα ε, κατακλειστεί από ευρωπαϊκά προϊόντα, γιατί θα πρέπει να δείτε και το καλάθι του, του ετηνισιακού νοικοκυριού. Νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου δημιουργεί ε, πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους ε, τινήσους εμπόρους που προσβλέπουν σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά που είναι η ευρωπαϊκή από ότι ο κίνδυνος που θα δημιουργηθεί από τον κατακλυσμό των ευρωπαϊκών προϊόντων στην Τινησία. Και φυσικά περιμένουμε αντίστοιχο άνοιγμα από την ευρωπαϊκή αγορά και μια αντίστοιχη υποστήριξη σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε λίγο μεγαλύτερη δυσκολία με το εμπόριο, διότι οι εμπορικέ μα ε, δραστηριότητε σήμερα στην Τινησία, ακόμη και στο εσωτερικό τη χώρα, δεν είναι αρκετά απελευθερωμένε. Ξεκινήσαμε με τον νόμο για τις επενδύσεις και αρχίσαμε να επιβάλλουμε μια προοδευτική απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών, διότι είχε αναπτυχθεί το παράλληλο εμπόριο, παράλληλη αγορά, εξαιτία του προστατευτισμού της ε, στεγανοποίησης της αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε το σωστό πέρασμα προς τον ανταγωνισμό, ε, την ανταγωνιστικότητα εντός χώρας. Βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα της όλης συζήτησης θα έχουμε στο πρώτο τρίμηνο την πρώτη σοβαρή αποτίμηση και νομίζω ότι ε, η προβλεπόμενη διάσκεψη θα είναι μια σημαντι... ένα σημαντικό βήμα. Η Λιβύη. Η Λιβύη είναι πράγματι ένα ποσοστό κινδύνου σοβαρό για μας. Βεβαίω όλα αυτά είναι λίγο τυχαία, αλλά έχουμε σοβαρό κίνδυνο σήμερα. Ξέρετε ότι το 2011 η Τινησία υποδέχτηκε 1,2 εκατομμύρια Λίβιους και ξένους πρόσφυγες στην επικράτειά μας και μας εξέπληξε η αντίδραση των ε, Τινήσεων στον Νότο οι οποίοι υποδέχτηκαν στα σπίτια τους τις οικογένειες των προσφύγων. Τους στήριξαν. Ήταν ε, υποδειγματική η συμπεριφορά τους και η στάση των ανθρώπων. Με πολύ μεγάλη διακριτικότητα όπως πρέπει. Ε, σήμερα φοβάμαι ότι αν προκύψει και άλλη κρίση και είναι και πιο σοβαρή στην Λιβύη, πράγμα που το φοβάμαι, η, την μόνη τη δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί. Δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πραγματικά δηλαδή ελπίζουμε ότι θα υπάρξει εδώ έντονη σαφή συνεργασία και στήριξη από την Ευρώπη. Για όσα θα συμβούν στη Λιβύη, για να προβλέψουμε, να προλάβουμε όσα μπορεί να συμβούν. Ελπίζουμε ότι η Λιβύη θα βρει τη σωστή ισορροπία με το ΙΝΟΙΕ και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθούν μας με τις γειτονικές χώρες να επηρεάσουν. Ε, αλλά εάν περάσουμε σε ένα σενάριο έστω και προσωρινό οξυμένης ε, έντασης στην Ευρώπη, ε, στην Λιβύη, συγγνώμη, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην Τινησία. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά. Διατηρούμε τις ελπίδες μας ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα, αλλά έχουμε και συνέστηση ότι πρέπει να γίνει δουλειά για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Θα κινητοποιηθούμε λοιπόν και έχουμε ήδη προχωρήσει. Έχουμε 220 χιλιόμετρα ε, χαντάκι που έχουν ε, σκάψει δικοί μας στρατιώτες ε, με τη δική σας βοήθεια και τεχνολογική στήριξη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη φύλαξη των συνόρων εγκαίρως σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη Λιβύη. Η Λιβύη κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοικοδομηθεί. Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για αυτά μπορεί να δουν την, την Ισία ως μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετήσει τη μελλοντική ανάπτυξη και τη δική μας βεβαίως και της Λιβύης ίσως. Ε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που το σχολιάζουμε όταν μιλάμε με τους εταίρους μας και τους υπόλοιπους συνεργάτες ε, σε επίπεδο διεθνών συνομιλητών, οι εταίροι μας ε, ανησυχούν. Επίπεδο χρέος 53% του ΑΕΠ, τα 2 τρίτα σε ξένο νόμισμα Έχουμε κάποιε δυσκολίε με το σωσίγιο πληρωμών λόγω τη πτώση του τουρισμού, 40% ε, λιγότερα έσοδα φέτο, αλλά έχουμε και τι θεμητέ προσδοκίε ότι η Τινησία ω προ την εξέβρεση τη οικονομική ισορροπία θα τα καταφέρει. Οι επενδυτέ ανησυχούν αν με τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα βεβαίω θα μπορέσουμε να πετύχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, διατηρώντα την απαραίτητη δημοσιονομική ισορροπία. Προφανώ ταυτόχρονα το Μάρσαλ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για να την πει κανείς έτσι εύκολα, αλλά ένα μίνι Μάρσαλ δεν θα μας πείραζε για να επιταχύνουμε την οικοδόμηση των απαραίτητων υποδομών είτε στο οικονομικό σύστημα είτε στο κοινωνικό και γι' αυτό χρειάζονται χρήματα. Πώς το χρήμα και πώς η Ευρώπη μπορούν να κάνουν περισσότερα. Η Ευρώπη είναι από τους πιο σημαντικούς ε, διάβλους ε, οι πηγές, για να το πω έτσι, ε, κονδυλίων. Όλοι βεβαίω θέλουν ένα τέτοιο εργαλείο βοήθεια όταν βρίσκονται σε δυσκολία. Μπορούμε να χρεωθούμε κι άλλα, αλλά προτιμούμε να μείνουμε στο 50-60%. Υπήρξατε ο πρώτο δωρητή ω Ευρωπαϊκή Ένωση στη βοήθεια που προσφέρθηκε στην Τινησία τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν χώρε που πήραν πολύ περισσότερο από εμά, 5 και 6 φορέ παραπάνω από εμεί, αλλά και άλλε χώρε που δεν έδωσαν τίποτα, ε, ιδίω χώρε του κόλπου. Ε, εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση τον Ιούνιο. Να πω ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτος μας εταίρος. Η Ευρώπη ε, πραγματικά συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και τον εξυγχρονισμό της Τινησίας. Και είναι ένας από τους πρώτους δωρητές. Με ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, με πολύ σαφείς στόχους και με συγκεκριμένη ε, στήριξη. Η ηλεκτρική διασύνδεση τη Ευρώπη με την Τινησία είναι επίση πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρο μα εξέφρασε τη στήριξή του προ αυτό το πρόγραμμα και ελπίζουμε να υλοποιηθεί. Να υπάρξει η διασύνδεση, διότι έχουμε γίνει ένα ε, Εισαγωγε... μια χώρα που εισάγει ενέργεια, το να παράγουμε ενέργεια θα είναι ένα τεστ πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες διασύνδεσης, γιατί έχουμε μεγάλη κατανάλωση το καλοκαίρι, εμείς αντιστρόφως από εσά. Αυτή την ιδέα που εξέφρασε και ο βουλευτής σας για ένα ειδικό ταμείο για την Τινησία μας, συγκεκριμένα ποσά στήριξης θα είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, Έχουμε μπροστά μας κάποιο χρόνο, αλλά μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσα έγιναν μεταξύ 2011-2015 εντωμεταξύ. Έχουν γίνει πολλά και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στην Ευρώπη για όσα έκανε και για όσα θα μπορούσε να κάνει τα ερχόμενα χρόνια. Αυτό που πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε είναι ότι αν επιτεθεί κανείς στην Τινησία, επιτίθεται στην Ευρώπη. Η εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την ευημερία είναι μια προσπάθεια που πρέπει να μοιραστεί η Ευρώπη με τις χώρες του Νότου. Είναι μια πολιτική πράξη υπέρ της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που μας περιγράψατε το φιλόδοξο σχέδιό σας, τη στρατηγική σας και κάποιες, που μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, και με αυτό ολοκληρώνουμε την ε, συζήτησή μας. Ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας σήμερα. Θα ξανασυνεδριάσουμε την ερχόμενη Δευτέρα 7 το βράδυ. Καλή σας μέρα και καλή όρεξη.